Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this meeting. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στην συνεδρίαση της επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Λάβατε όλη την ατζέντα, υποθέτω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια επ' αυτής. Αφού λοιπόν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Βλέπετε στο Κόκομπου Info, στο φυλάδιο τι γλώσσες έχουμε σήμερα. Ε, μεταδίδεται από το ίντερνετ τη συνεδρίαση. Όπως συνήθως, να περάσω στο 3 της ημερήσιας ε, διάταξης. Διορισμός 8 μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Την πρώτη ώρα θα ακούσουμε τα τρία μέλη, τα οποία ήδη αποτελούν μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του παρόντος και μιλάμε για ανανέωση της σύμβασης. Θα πρότεινα καθίσει εξ αυτών να μιλήσει επί 5 λεπτά και στη συνέχεια οποιοδήποτε βουλευτής μπορεί να θέσει ερωτήσεις τις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν και αν υπάρχει χρόνος θα γίνουν και συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ιδάλλως, αν συμφωνείτε, να δώσω το λόγο στον κύριο Πίνξτεν για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω όλη την ώρα στην μητρική μου γλώσσα, αλλά ξέρετε ότι στη χώρα αυτή το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ik zei Είπα λοιπόν σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας μου στην μητρική μου γλώσσα. Μιλώ α, μόνο λίγο τη γλώσσα μου, γιατί και εσείς Πρόεδρε την ίδια γλώσσα μιλάτε και επειδή θα γνωρίζετε ότι το να μιλά κανείς τη δική του γλώσσα στην ε, χώρα αυτή αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα από σεβασμό λοιπόν προς την κοινότητά μου. Θα πω δύο λόγια στη μητρική μου γλώσσα, στα Ολλανδικά. Αυτό που καταρχάς θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής και αυτό το κάνω το εκφράζω προς τους βουλευτές που βρίσκονται εδώ σήμερα το πρωί. Ξέρετε ότι γνωρίζω πολύ καλά το κοινοβουλευτικό γίγνεσθε και γνωρίζω το, το κοινοβουλευτικό γίγνεσθε και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και καταλαβαίνω ότι οι βουλευτές δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω ότι έχουν παράλληλες υποχρεώσεις, τρεις, τέσσερις και πέντε καμιά φορά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο για την άριστη συνεργασία με το Ελεκτικό Συνέδριο και με την Επιτροπή σας. Αυτό λοιπόν καταρχά, Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να στραφώ εν συντομία. στο συνοπτικό σημείωμα το οποίο σας διαβίβασα. Όταν ε, ε, διορίστηκα στο Ελεκτικό Συνεδρίο πριν από έξι χρόνια, ήμουν μέλος της ομάδας Τώρα είμαι στην τρίτη αίθουσα, στο τρίτο τμήμα και είμαστε υπεύθυνοι για εξωτερικές δράσεις. Γιατί λοιπόν διορίστηκα στην τρίτη ενότητα, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ο προκατοχός μου ήταν πάντα σε αυτό το τμήμα και ίσως αυτό να αποτέλεσε το λόγο. Αυτό μου επέτρεψε να καταρτήσω μία σειρά εγγράφων κατήρθησα πέντε εξειδικευμένες εκθέσεις με όλη τη μετριοφροσύνη θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός αριθμός τέτοιων ειδικών εκθέσεων γιατί ξέρετε ότι μία ήταν για το τσουνάμι προετοιμάσαμε και μία έκθεση follow-up Στη συνέχεια, τρία χρόνια αργότερα, προετοίμασα μια έκθεση επίσης για τον τυφώνα Μέιτς και το τσουνάμι και τις σχετικές εργασίες αποκατάστασης. Επίσης ε, για τον ΟΙΑ μία έκθεση την οποία ολοκλήρωσα φέτος για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που ε, διοχετεύονται μέσω του ΟΗΕ. Αυτές λοιπόν είναι οι πέντε εξειδικευμένες εκθέσεις τις οποίες προετοίμασα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Επίσης συνέβαλα για το κεφάλαιο στο κεφάλαιο για το 2006 και το 2007 και χαίρομαι που από τις αρχές του έτους οι συνάδελφοι από το τμήμα 3 με διόρισαν, με επέλεξαν, δεν ήταν πραγματικές εκλογές, για να, είμαι, για να καταστώ ο πρόεδρος του τμήματος 3. Συμμετέχω λοιπόν και στην Διοικητική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο πρόεδρός μας. Η Διοικητική Επιτροπή, πώς να το θέσω, αποτελεί, αν θέλετε, ε, ένα προκαταρτικό σχήμα μιας Διοικητικής Επιτροπής. Θα, κλείνω, θα κλείσω λοιπόν με τα τρία αυτά σημεία, Πρόεδρε. Ποιοι είναι οι στόχοι μου. Καταρχάς, θέλω να συμβάλλω στην διατήρηση υψηλών προτύπων για το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο, γιατί δεν είναι μια ομάδα δημοσιογράφων με κάθε σεβασμό, αλλά θα πρέπει να δουλεύει με εντελεχή τρόπο. Κατά δεύτερον, να προωθήσω τις καλές ε, σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εκπροσωπείται τον ευρωπαϊκό φορολογούμενο και εμεί για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο εργαζόμαστε. Είναι άρα πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλές εργασιακέ σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τους άλλους εμπλεκομένους φορείς. Νομίζω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διαφορά με τις εκθέσεις μας και θα ήθελα, αν μου δοθεί η ευκαιρία, να πω δύο λόγια παραπάνω στο σημείο αυτό. Πιο μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος κύριε Πίνγκστεν και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Καλτέρα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Ήταν τιμή για μένα και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη να υπηρετήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λογικό Συνέδριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας ως υποψήφιος για το Ελεκτικό Συνέδριο και από το Μάρτιο 2000 όταν έγινα μέλος για πρώτη φορά όταν υποψήφισε πρώτη φορά προσπάθησα με τις προσπάθειές μου να επιτρέψω στο σώμα των ελεκτών να υλοποιήσει την αποστολή του στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν 10 χρόνια λοιπόν είμαι υπεύθυνο για τις τραπεζικές δραστηριότητες και για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2002 έγινα μέλος της ΔΑΣ και είχα την χαρά και την ευχαρίστηση να συνεργαστώ με διάφορα μέλη της Επιτροπής σας και ήμουν εισηγητής για τον ενιαίο έλεγχο στο λεκτικό συνέδριο. Κάτι που ακολούθησε αργότερα ως έκθεση, ως κατευθυντής γραμμές και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Κομισιόν και το οποίο βλέπουμε να τα αγκλάται σήμερα και στις χρηματοοικονομικές προοπτικές και στους κανονισμούς. Όταν ξεκίνησα το 2006 την τρίτη μου θητεία ήμουν στην οριζόντια ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό και τις μεθόδους αξιολόγησης ήμουν υπεύθυνο τότε για τις μεθόδους ανάπτυξης μεθόδων ελέγχου ποιότητας. Το 2008 εξελέγει πρόεδρος για τρία χρόνια και μετά επανεκλέχτηκα. Στην πρώτη μου θητεία ως πρόεδρος το ελεκτικό συνέδριο ολοκλήρωσε μια εσωτερική διαδικασία αναθεώρησης κάτι το οποίο επέτρεψε στο σώμα μας να αναθεωρήσει τους εσωτερικούς κανόνες, να θεσπίσει το σύστημα με τα τμήματα και να αναπτύξει μια διαδικασία που ανέφερε και ο κύριος Πίξεν ως ε, βελτίωση της εσωτερικής διοίκησης. Ως τμήμα αυτής της διαδικασίας υιοθέτησε το λεκτικό συνέδριο και μια στρατηγική ελέγχου που απέβλεπε στη βελτίωση της ποιότητας της δουλειά μας και των αποτελεσμάτων της ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σε συνεργασία με την Επιτροπή σας. Επίσης, το συνέδριο μπόρεσε να συνεισφέρει ενεργά στις δημόσιες συζητήσεις για την αναθεώρηση για τους δημόσιους ε, διαγωνισμούς και την ε, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της ε, δράσης του ελεκτικού συνεδρίου χρησιμοποιώντας καλύτερα τους πόρους που ήταν στη διάθεσή του. Και αυτό ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχα στην πρώτη μου θητεία ως πρόεδρος και το διατήρησα ως προτεραιότητα για το μέλλον. Και από την έννοια αυτή, αν ανοηθεί η θητεία μου και έχω την εμπιστοσύνη της Επιτροπής σας, θα προσπαθήσω να αναπτύξω μια νέα εξωστρεφή πολιτική για το συνέδριο που θα επικεντρώνεται στην εντατικοποίηση των επαφών του συνεδρίου με τους διάφορους εμπλεκόμενους ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Μετά θα χρησιμοποιούσα καλύτερα του εσωτερικού κανόνε ώστε να βελτιστοποιήσουμε του πόρου που έχουμε ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί. Και τρίτον, θα προσπαθήσω να προωθήσω την δημόσια λογοδοσία στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του εθνικού οργανισμού μαζί με τα ελεκτικά συνέδρια βέβαια και των χωρών μελών. Επίσης, Θα προσπαθήσω να διαδώσω περισσότερο το μήνυμά μας ώστε να έχουμε περισσότερο αντίκτυπο ως δράση του ελεκτικού συνέδριου. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να συμβάλλω θετικά στην βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των ευρωπαϊκών οικονομικών, δημοσίων οικονομικών και θα ήθελα το Ελεκτικό Συνέδριο να δραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεξάρτητο όργανο με επαγγελματικότητα που συμβάλλει σε όλες τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ που μου δίδετε την ευκαιρία να βρεθώ εδώ σήμερα και να ζητήσω την εμπιστοσύνη σας για τη δεύτερη μου θητεία ως μέλος της, της... του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Όπως ξέρετε, διοριστικά τον Ιούνιο φέτος, αντικαθιστώντας τον προκάτοχό μου στο Ελεκτικό Συνέδριο και όπως είπα, στην συνοπτική παρουσίαση του βιογραφικού μου που σας έστειλα, είμαι μέλος του τρίτου τμήματος που είναι υπεύθυνο για τις εξωτερικές δράσεις και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αμέσως για την ετήσια έκθεση που αφορά τι εξωτερικές δράσει και την διεύρυνση. Ήμουν υπεύθυνο για την απαλλαγή που θα συστήθω εδώ στην Επιτροπή σα τον Γενάρη. Ταυτόχρονα ήμουν υπεύθυνο για τρει διαδικασίε ελέγχου. Η πρώτη, η οποία βρίσκεται στη δικασία διασταύρωση και αφορά την τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της επιστημιστικής βοήθειας στην υποσαχάρια Αφρική. Η δεύτερη διαδικασία για την οποία είμαι υπεύθυνο και η οποία ολοκληρώνεται μέσω προκατακτικής μελέτης αφορά την διαχείριση της Κομισιόν όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια στα ευαίσθητα κράτη όπως λέγονται και η τρίτη δουλειά θα ξεκινήσει του χρόνου και αφορά την ε, αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αν δούμε τα θέματα οριζόντιας συζήτηση του συνεδρίου, εγώ συμμετέχω στην, προετοιμασία της επόμενης στρατηγικής του συνεδρίου που επικοινωνούνται ιδιαίτερα στα θέματα αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να συμβάλλω στην απλούστευση των διαδικασιών και να παράσχω μια πιο επικεντρωμένη προσέγγιση με μελέτης. Ως μέλος του συνεδρίου έχω την ευθύνη να διασφαλίσω την συμβολή μου στην ε, αρρωγή στην Επιτροπή σας, όχι μόνο βεβαίως παρέχοντας έγκαιρα τις απαραίτητες εκθέσεις, αλλά επικεντρώνοντας τη συζήτηση για τα κύρια θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θεωρώ ότι ο ρόλος της Επιτροπής σας είναι κύριος όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του στόχου. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. And Ευχαριστώ κύριε Βέσπερκ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη και καταρχήν στην εισηγήτριά μας. Ε, αν θέλετε να πείτε τίποτα. Sí. <clears throat> Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους τρεις υποψηφίους για την παρουσία τους και την υποψηφιότητά τους για ανανέωση της θητεία τους. Καταρχήν για τον κύριο Πίντσεν θα ήθελα να το ρωτήσω για την εργασία του σε αυτήν την πρώτη φάση στο Ελεκτικό Συνεδρίο εργάστηκε κυρίως στον τομέα των εξωτερικών δράσεων Θα ήθελα να το ρωτήσω λοιπόν το εξή. Ανέκαθεν είχαμε προβλήματα με τα προγράμματα που αφορούν συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ιδιαίτερα στα πλαίσια του ΟΗΕ. Θα ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Νομίζετε ότι με τις ειδικέ εκθέσεις και με την αφοσίωσή σας ως κοσμήτορα του τρίτου τμήματος θεωρείτε ότι οι δράσεις αυτές έχουν βελτιωθεί ή με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βελτιωθούν γιατί στις τελευταίες συζητήσει που είχαμε για τη συνεργασία και την διαφάνεια των πόρων του ΟΗΕ και ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη και τη δική μα χρηματοδότηση, τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφή. Και ξέρω ότι εργαστήκατε επίση και στην Επιτροπή που ασχολήθηκε με τα θέματα της Europol, ένας φάκελος αρκετά περίπλοκος που παραμένει σε κρεμότητα. Θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στην Κοινή Επιτροπή για την Europol συνέβαλε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να βρεθεί μια διέξοδο σε αυτό το πρόβλημα. Και εσείς είπατε στο τέλος ότι οι στόχοι σας για μια μελλοντική θητεία περιλαμβάνουν τη βελτίωση των διαδικασιών μέσω της βελτίωσης των εκθέσεων. Θα μπορούσατε να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα μπορούσατε να κάνετε ώστε να βελτιωθούν αυτές οι συγκεκριμένες εκθέσεις. Ευχαριστώ. Mr. Κύριε Πίξον, μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντως ε, εργάστηκα πάνω στην συνεργασία ε, με το web και αρχικά τα είχα συμπεριλάβει όλα αυτά σε μία εισήγηση. Μετά όμως σκέφτηκα ότι το θέμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήξερα ότι και το Κοινοβούλιο εργαζόταν πάνω στο ίδιο θέμα, οπότε ε, έφτιαξα δύο ξεχωριστές εκθέσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα είπα στην εισήγηση, απλώς θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα και ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι μπορώ να μιλήσω ε, για τον εαυτό μου λέγοντας ότι θέλω να τονίσω ότι είναι πιο ενδιαφέρον ενδεχόμενα για τα μέλη. Αυτό να, μόνο να πω. Πρώτον, ε, πρέπει να τονίσω ότι η νέα Κομισιόν μας έδωσε ε, μια επιλογή οργάνου, κάτι το οποίο είναι καινούριο και σε μένα ακόμα δεν είναι σαφές μετά από την προσφορά αυτή γιατί στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ε, ε, επέλεξε να δουλέψει με, το, ε, με τον ΟΙΕ και στη μία περίπτωση και όχι στην άλλη. Η, είχε το καθήκον να είναι δίκαιη η Επιτροπή και βεβαίως μπορεί να είχε πάρα πολύ ε, ισχυρούς λόγους να δουλέψει με τον ΟΗΕ αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να τους εξηγήσει αυτούς τους λόγους στο Κοινοβούλιο, το οποίο είχε κάνει πάρα πολλά. Στο μέλλον φαντάζομαι ότι θα ακολουθηθεί αυτή η πρακτική. Τουλάχιστον έτσι μου είπε ε, ο πρόσωπος της Επιτροπής τρεις εβδομάδες πριν. Δηλαδή η επιλογή ανάμεσα στα διάφορα όργανα θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη και από χρηματοοικονομική άποψη αλλά και από πολιτική και άλλες απόψεις. Ας σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα Είχαμε χτες τη συνεδρίασή μας ε, τις, ε, τα αποτελέσματα μιας, ε, ενός ελέγχου που κάναμε στο Λονδίνο και ένα μέρος του ελέγχου αυτού είχε γίνει με ε, με, το, με UNDP. Γιατί είπε, ρώτησε η Επιτροπή τι λόγος υπάρχει για, για αυτή την επιλογή. Καταρχήν είπαμε ότι υπάρχει, είναι μέσα στην Ένωση, ε, πρέπει να μπορεί να αποσταλεί μια αντιπροσωπεία. Στην ε, Βόρεια Κύπρο δεν μπορεί να αποσταλεί μια αντιπροσωπεία και δόθηκαν όλες αυτές οι εξηγήσει. Ε, και με αυτή την ανταλλαγή απόψεων που ήταν ικανοποιητική με την Επιτροπή είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι και πιστεύουμε ότι στο μέλλον έτσι πρέπει να δράσουμε για όλα τα εργαλεία, τα όργανα που χρησιμοποιούμε εφαρμογής. Ύστερα, το δεύτερον, ξέρουμε όλοι ότι ο ΙΕ είναι μια τεράστια οικογένεια ε, σε διάφορα θεσμικά όργανα του κόσμου ολόκληρου, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετικές δραστηριότητες ε, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που ασχολείται με διάφορα θέματα παγκοσμίως. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και να μην γενικεύουμε. Εγώ είδα μαζί με τους υπαλλήλους μου ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και μια πολύ καλή θετική σχέση με τον ΟΗΕ. Αν όμως χρησιμοποιήσει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ο ΟΗΕ, πιστεύω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να του ζητήσουμε είναι να μας πει πώς δαπανούνται αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα ε, πρέπει οπωσδήποτε, ο, εφόσον γίνεται η δαπάνη από τον ΟΗΕ να δίνεται μια εξήγηση και μια δικαιολόγηση. Ενώ δεν υπήρχε καν η αναφορά, μα καθόλου. Και αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Πρέπει, πιστεύω, ε, να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από αυτόν τον έλεγχο που ασκεί το ελεγκτικό συνέδριο να ασκήσει και πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι και το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ βασικό να πιέσει από αυτού του θέματος. Μήπως ε, για λόγους δημοκρατίας θα μπορούσατε να συντομεύετε. Ε, σας παρακαλώ πολύ κύριε Πίγκστεν. Ε, έχω πάρα πολλά να πω για τους διάφορους οργανισμούς, για... έμαθα πάρα πολλά από αυτόν τον έλεγχο. Αυτό που έμαθα ήταν ότι συνήθως θεωρούσαμε όλους τους οργανισμούς, τους επιμέρους του, του, του ΟΗΕ ότι ήταν ίσοι. Ε, όμως Υπάρχουν άλλοι που εφαρμόζουν, ορισμένοι που εφαρμόζουν τον κανονισμό πολύ πιο εύκολα, με μεγάλη ευχέρεια και άλλοι όχι. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ε, ε, έχουν διαφορετική θέση και ως προς τα, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μιλήσατε πολύ περισσότερο από τον προλαλήσαντά σας και θα συνεχίσουμε με τους επόμενους και το τελευταίο δεν θα το θέσουμε τώρα Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η εισηγήτρια θέλει να σας θέσει ερωτήματα. Θα ήθελα να κρατήσουμε, να τηρήσουμε το χρόνο ομιλία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο λεπτά για τις ερωτήσεις και δύο λεπτά για τις απαντήσεις. Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να... Ναι, Πρόεδρε, το κατανοώ αυτό. Και εγώ θα ήθελα να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Για τον κύριο Καλντέιρα να πω ότι τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε την παρουσία του, την προεδρία του και νομίζω ότι όντω υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην αντίληψη του ελεκτικού συνεδρίου ως αποτελεσματικό εργαλείο σε σχέση με το παρελθόν όπου αποτελούσε έτσι κάτι το απροσδιορίστο με συχνέ αρνητικέ εκπλήξει. Να ρωτήσω το εξή. Τα τέσσερα σε μια επανακοίνωση και παρουσίαση ω μελλοντικέ κατευθυντήρε γραμμέ σε σχέση με τι νέε αρμοδιότητε που συνοδεύουν του νέου μηχανισμού χρηματοδότηση και διάφορου άλλου μηχανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου εμπλέκεται ο Ευρωπαϊκό ο κοινωνικός περιπολογισμός, να το ρωτήσω το εξή. Δεν θα έπρεπε, και γνωρίζω ότι το κάνετε από την αρχή, επειδή αναδιονοργανώσατε σε μια πρώτη φάση το ελεκτικό συνέδριο. Δεν θα έπρεπε όμω να προβλέψουμε μια νέα δομή ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια, ακόμα και με τα περιφερειακά. Γιατί ε, θα βρεθούμε σε μια νέα δυναμική μετά από αυτή τη φάση. Και, στην, και για την επικοινωνία λέτε ότι θέλετε να βελτιώσουμε την επικοινωνία, να φτάσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στους πολίτες. Να μας πείτε αν έχετε συγκεκριμένες ιδέες από αυτού και κατά πόσο η βελτίωση της σχέσης με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια θα βελτιώσει και τη σχέση με το Συμβούλιο όσον αφορά την διαχείριση του κοινωτικού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και όλοι οι μηχανισμοί ε, τους οποίους ε, χρησιμοποιούμε στην παρούσα, στη νέα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο ολόκληρο εξάλλου για να αντιμετωπιστεί η χρηματοοικονομική κρίση. Όλα αυτά απαιτούν νέα όργανα και την παρέμβαση διαφόρων οργανισμών που πρέπει να αναλάβουν δράση. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, έχουμε ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα και ε, επιλέγουμε συνήθως τα όργανα τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά. Ε, τον σταθεροποιητικό ευρωπαϊκό μηχανισμό ε, που αφορά τις εγγύσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ένας έλεγχος από, τους, από, το, από το ελεγκτικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση του χρέους, την ευρωπαϊκή διευκόλυνση του χρέους, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια του σταθεροποιητικού ευρωπαϊκού μηχανισμού στο μέλλον, περνώντας μέσα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να λειτουργεί σωστά. Υπάρχει επίσης ένας ε, έλεγχος με ε, μια επιτροπή πέντα μελή Τρία από αυτά τα μέλη ανήκουν σε διεθνείς ε, οργανισμούς και ένα μέλος ανήκει υποχρεωτικά στο Ελεγκτικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Ε, συνεργαζόμαστε με τα εθνικά Ινστιτούτα, με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια πολύ στενά και ήδη ενσωματώσαμε τα αποτελέσματα συνεργασίας, κοινή εργασίας που είχαμε με την τσεχική ε, δημοκρατία σε θέματα γεωργίας και με τις ε, κάτω χώρες. Βεβαίως πρέπει κανείς να εξετάσει την ανάλυση κόστους-οφέλους και πιστεύω ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα στο να συνεργαστούμε σε αυτόν τον τομέα, να υπάρχουν δύο task ε, forces και για να δούμε τι ε, εργασία μπορούμε να, επιτελέσουμε στον τομέα της φορολογικής ε, πολιτικής με τα νέα δεδομένα, τα οικονομικά των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών που εμφανίζονται σιγά σιγά. Ε, και πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχουν σχέση με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής και τα σχετικά φορολογικά σχέδια πρέπει να ειδωθούν πιο αναλυτικά. Αυτή είναι η εργασία που επιτέλεσα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε και άλλες ερωτήσεις ε, κυρία εισηγήτρια. Όχι. Ωραία. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκρίς. Κύριε Κρέτσλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ήθελα να θέσω την ερώτηση προς όλους τους υποψηφίους. Αν υπήρξαν κατά την προηγούμενη θητεία τους ε, ε, περιστάσεις όπου έπρεπε να προστατεύσουν ένα κράτος μέλος και ποιες ήταν αυτές οι περιστάσεις. Κατά δεύτερα, να ρωτήσω καταρχά τον πρόεδρο Καϊτέιρα. Υπάρχει ε, μια μεταβίβαση περίπτωσης του από την Όλαφ στο ελεγκτικό συνέδριο για απάτη. Αληθεύει ότι το ελεγκτικό συνέδριο αναλαμβάνει τα δικηγορικά έξοδα για το εμπλεκόμενο άτομο, άρα δηλαδή τα διοχετεύει ουσιαστικά στον φορολογούμενο. Και ποια είναι η αιτιολόγηση αν αυτό ισχύει. Γιατί ο φυσιολογικός, κανονικός πολίτης που μαθαίνει κάτι τέτοιο δεν ε, αρέσκεται και δικαίω σε αυτά τα φαινόμενα. Μία άλλη ε, ερώτηση. Ασκήσαμε ιδιαίτερη κριτική στις εξειδικευμένες εκθέσεις γιατί δεν ε, περιλαμβάνουν αυτά που χρειαζόμαστε για να δράσουμε. Δηλαδή μια σαφή εξήγηση του που ε, έγινε το πρόβλημα. Θεωρώ ότι εξακολουθούν να είναι υπερβολικά γενικόλογες αυτές οι εκθέσεις και μέσω του είδους ε, εργασία στο Ελληνικό Συνέδριο είναι έτσι. Τι θα επιχειρήσετε να κάνετε προκειμένου να μας ε, διαβιβάζετε καλύτερες ε, εξειδικευμένες εκθέσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εγώ έχω ασχοληθεί με πολλές εξ αυτών και διαπιστώνω πάντα τέτοιες αδυναμίες. Θα συνεργαζόσασταν στα πλαίσια μια τέτοια ανάλυσης για την αποτελεσματικότητα από πλευράς διοργανωτική του ηλεκτρικού συνεδρίου προκειμένου να αλλάξει κάτι σε αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι η ερώτηση ήταν προς όλους τους υποψηφίους. Δεν ξέρω, θέλετε να ξεκινήσετε. Κύριε και δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση αν σωστά την ερμηνεύω. Αν είχα κάποιο λόγο να προστατεύσω το, τη χώρα μου. Όχι, είναι η απάντηση και του πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Μετά θέσατε μία ερώτηση για τις ειδικέ εκθέσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να εξελιχθούν, να μεταξελιχθούν οι ειδικέ εκθέσεις από την σύντομη σχετικά εμπειρία μου, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που είναι πιο ενδιαφέροντες από ότι Καταρχάς, λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε θέματα εστίασης. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προετοιμάζω στην παρούσα φάση μια προκαταρτική έκθεση για την έκθεση για τα ευαίσθητα κράτη. Θεωρώ ότι είναι πολύ περιορισμένη και εις βάθος η ανάλυση μου. Θεωρώ ότι θα ήταν κακοφόρο και υποφελές να προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε έτσι να εργαστούμε. Αυτό σκοπεύω να κάνω πάντως. Τώρα το θέμα της εγκυρότητας. Κοιτάξτε, ποτέ δεν μπορούμε να περιορίσουμε ή να κάνουμε συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα, γιατί αν ε, συμβεί αυτό δεν θα είναι ενδιαφέρον το υλικό. Αλλά ενδεχομένως να μπορέσουμε να μπορούσαμε να προβλέψουμε κάποια μηχανισμό ταχείας αντίδρασης ε, σε ό,τι αφορά τέτοιες εκθέσεις πιο σύντομες από τους 18 μήνες που προβλέπονται τώρα. Αυτό θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Πίγκστεν. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Για την πρώτη ερώτηση. Ποτέ δεν έχει προσογήσει κανείς για κάποιο βελγικό θέμα. Ποτέ δεν έχω ζητήσει εγώ ίδιος βελγικό φάκελο και δεν έχω δει ποτέ βελγική υπόθεση. Και αν κάποιος με προσέγγιζε θα έλεγα ότι όχι δεν ενδιαφέρομαι. Είναι αδιανόητο ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Για παράδειγμα, όταν ε, υπάρχει εντολή για συναλλαγές, ε, είναι αδιανόητο να επηρεαστεί από οποιαδήποτε ε, πλευρά. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτό μπορώ να σας το πω. Δεύτερη ερώτηση, πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Να σα πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι ειδικέ αυτέ εκθέσει. Καταρχά, θα πρέπει να είναι σύντομε, γρήγορε και πολύ συγκεκριμένε. Η έκθεση για το τσουνάμι. Θεωρώ ότι ήρθε στη σωστή χρονική στιγμή. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν είναι εύκολο αυτό αν, αν θέλουμε να γίνει έλεγχο για την υπηρεσία εξωτερική δράση, να το ξεκινήσουμε τώρα. Τι θα γίνει, θα περιμένουμε να εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τέλου. Δεν είναι πάντα εύκολο λοιπόν αυτό. Το μήνυμα είναι ότι δεν είμαι υπέρ ένα μήνυμα με ελεγκτικού όρου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μεταφράζουμε, να ερμηνεύουμε τα μηνύματα που αποστέλουμε. Γιατί θα πρέπει να είναι κατανοητά και στον Ευρωβουλευτή και στον Ευρωπαίο πολίτη. Αν στην Αμερική ο Υπουργό ε, Οικονομικών μπορεί να γράφει άρθρα σε εφημερίδε στου Financial Times κάθε δύο εβδομάδε και εμεί το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, Λέει και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να απαντήσω στα ερωτήματα της κυρίας Γκρέσλε. Καταρχάς, νομίζω ότι τα 11 χρόνια που έχω ε, εργαστεί στο ελεγκτικό συνέδριο, νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι είμαι αμερόληπτος, ε, άρα ασφαλώς και απαντώ αρνητικά στο πρώτο ερώτημα. Αναφερθήκατε στις ειδικές εκτέσεις. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας σύνδεσμος, μια σύνδεση με το θέμα της επικοινωνίας που είχε θέσει ως ερώτηση η κυρία Γιάλα Σάντρη και δεν απάντησα. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση τις ειδικές εκθέσεις να τις καταπτύσσουμε πιο γρήγορα με ουσία ισοσκελίζοντας ε, θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας με μία γλώσσα κατανοητή από εσά εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και από τους πολίτες. Αυτό προσπαθούμε να αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή μας. Φυσικά, ε, τις εκθέσεις ε, της διαβάσης του Συνέδριου. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε καν να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που τίθενται και αυτό δεν προωθεί το πνεύμα της επικοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε νέα αποτελέσματα τα οποία θα ανταποκρίνονται με καλύτερο τρόπο στις ανάγκες του Κοινοβουλίου, στις συστάσεις σας. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δράσουμε ενεργά για να βρούμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται προκειμένου να πετύχουμε ακριβώς αυτός που αναφέρθηκε στοχευμένα, γρήγορα, ποιοτικά αποτελέσματα με σεβασμό των προδιαγραφών ε, και τις μεθοδολογίες που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο επαγγελματικός έλεγχος. Για την όλα τώρα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ξεκίνησε πριν από ένα έτος και είμαστε... έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Όλαφ και στα αποτελέσματα. Αλλά σύμφωνα με το καταστατικό κανονισμό για το προσωπικό, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν ένα θεσμικό όργανο να τους ε, συνδράμει σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά έχουν ε, διαβιβαστεί και στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου για να γίνει ποινική έρευνα και μετά από αυτά το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να καταγγείλει όλες τις συμβάσεις ως προς την ασφάλεια με εξωτερικούς παρόχους. Και με το μέτρο αυτό το ελεγκτικό συνέδριο έκανε εξοικονόμηση σημαντικών κονδυλίων από τον προϋπολογισμό. 6.000 ευρώ ανά έτος. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν ακολούθησε πολύ απλά τους κανόνες του κανονισμού που προβλέπουν προστασία των υπαλλήλων και κατά δεύτερον το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να παρέχει στοιχεία στην Όλαφ και θα το πράξει αυτό και τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αλλά είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι θα λάμψει η, η αλήθεια στο θέμα αυτό. Σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα γιατί έχουμε τρεις βουλευτές που θέλουν να θέσουν ακόμα ερωτήσεις. Να προτείνω να ακούσουμε τους τρεις βουλευτές και τις ερωτήσεις τους. Δύο λεπτά ο καθένας και μετά να απαντήσουν οι τρεις υποψήφοι και τέλος θα μπορέσει η συγκήτρια να κάνει μια σύνοψη. κυρία Ιβρακοβά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συγκήτρια έθεσε ήδη την ερώτηση, αλλά να επανέλθω στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι σημαντικό αυτό για την εκπομπή μας γιατί ξεκινήσαμε μια ξεχωριστή μελέτη για το ρόλο των χρηματοοικονομικών εργαλείων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού και κύριε Καλτέρα είπατε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας με 60 δισεκατομμύρια ευρώ θα παρακολουθείτε από το συνέδριο. Τι γίνεται όμως με το ESM. Ξέρουμε ότι το 2013 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα αντικαταστήσει τα δύο εργαλεία τα οποία είναι προσωρινά και ένα τμήμα των 60 δις θα διαιρεθεί στο ESM. Πώς θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία το λεκτικό συνέδριο. Ξέρω ότι λέει κάποια πράγματα συνθήκη, αλλά μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ώστε ότι εσείς θα κάνετε ε, ό,τι μπορείτε ώστε να διασφαλιστεί ένας ενεργός ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κάλβιν παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καλτέρα. Αλλά να πω προηγουμένω ότι δούλεψα με τον κύριο Πίντσεν για, το θέμα της αποκέντρωσης εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω... είχα μια καλή συνεργασία μαζί του. Ερώτηση πάντως για τον κύριο Καλτέρα. Ο έλεγχος και η άσκηση του ελέγχου αποτελεί ένα επάγγελμα που ρυθμίζεται. Και εγώ είμαι μέλος στο Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Ελεκτών και έχουμε μέλη με τελείως διαφορετικό υπόβαθρο και τελείως διαφορετικά, διαφορετικές προδιαγραφές επαγγελματικέ. Ο έλεγχος δεν είναι πολιτική πράξη, την πολιτική την ασκεί ένα όργανο όπως το Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι στο επιμελητήριο των Ευρωπαίων Ελεκτών θα έπρεπε να ισχύουν κάποιες ελάχιστε προδιαγραφές. Έχετε πρόθεση να προτείνετε κάποιες ελάχιστε προδιαγραφές για τους Ευρωπαίους ελεκτές ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκόντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επεκτείνοντας την ερώτηση του συναδελφού, να πω ότι φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει ένα κώδικα διοντολογίας που αφορά τα παγκόσμια όργανα ελέγχου λογαριασμών. Υπάρχουν λοιπόν δύο θέματα που θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Σύγκρουση συμφερόντων. Όταν ανέκυψαν τέτοιες περιπτώσεις, πώς τις λύσατε. Δεύτερον, για τις αρμοδιότητες στα πλαίσια του κώδικα Διοντολογία. Έχετε κάποια κατάρτιση συνεχόμενη, κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλου του ελεκτέ. και τι ακριβώ προτείνεται ω κατάρτιση στα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση προ τον κύριο Βεσμπέργκ. Η συνθήκη λέει ότι για ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να έχουμε μία από τις δύο προϋποθέσεις ή συνθήκες είτε να είναι κανεί μέλο του Εθνικού ελεκτρικού Συνεδρίου ή να έχει ιδιαίτερη κατάρτιση όσον αφορά τον έλεγχο. Βλέποντα λοιπόν το βιογραφικό σα, δεν κατάλαβα ακριβώ ποια είναι η φύση των ιδιαίτερων προσόντων που έχετε εσεί όσον αφορά την άσκηση του ελέγχου στα πλαίσια πάντα τη υποψηφιότητά σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η πρώτη ερώτηση, αν κατάλαβα καλά, απευθύνεται στον κύριο Καλτέρα. Η δεύτερη στον κύριο Πίκτσεντ. Όχι, διορθώνουν οι προλαλήσαντε. Δεν είναι έτσι, Πρόεδρε. Τέλο πάντων, λέω πρώτα θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Καλτέρα να, να απαντήσει στα ερωτήματα. Πρόεδρε. Δύο λεπτά να απαντήσω. Γι' αυτό που είπε η κυρία Ιβακόβα. συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια μέσω και της Επιτροπής Επαφής ώστε να διασφαλιστεί ο καταλληλότερος έλεγχος και υποπτία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Βεβαίως, Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο είναι ο ελεκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων. Υπάρχει λοιπόν ο ρόλος της Ένωσης σε αυτούς τους μηχανισμούς σταθερότητας, οπότε αυτός ο ρόλος αναπόκειται κυρίως στο Ελεκτικό Συνέδριο. Και οτιδήποτε εκτίθεται ή σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό προπολογισμό παρακολουθείται και υποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτή είναι η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα για τον κύριο Κάλβιν. Για τα προσωπικά κριτήρια και προδιαγραφέ για το επιμελητήριο. Να κάνω δύο σχόλια. Καταρχήν, το διαφορετικό υπόβαθρο των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου κάτι από μόνο του, νομίζω ότι αποτελεί ένα παράγοντα που εμπλουτίζει το όργανο, γιατί μπορεί κανείς να αποφεληθεί από την τεχνογνωσία, που έχουν ακαδημαϊκοί, που έχουν μέλη των ε, Δυτικών Συμβουλίων Κεντρικών Τραπεζών σε χώρες μέλη που έχουν υπάλληλοι όπως εγώ. Νομίζω ότι αυτό εμπλουτίζει το όργανο. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος ακόμα και περιθώριο για τις χώρες μέλη ώστε να, να εντοπίσουν τους καταλληλότερους υποψηφίους σύμφωνα με τα κριτήρια των συνθήκων. Αν η συνθήκη λέει ας πούμε όπως στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι το Συμβούλιο κάνει ακρόαση για τους υποψηφίους και εξετάζει το βιογραφικό τους Αυτή η εξέταση γίνεται από ακαδημαϊκούς, από πρώην μέλη του δικαστηρίου κλπ. κλπ από μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και λοιπά. Αυτό επιτρέπει στο να αξιολογήσουμε καλύτερα και για τον κώδικα διοντολογίας. Νομίζω ότι υιοθετήσαμε ένα ενημερωμένο κώδικα διοντολογικό για όλα τα μέλη του προσωπικού και αυτός ο κώδικας προβλέπει τα απαραίτητα για την ρύθμιση σύγκρουσης συμφερόντων. Ακολουθούμε όμως τον παραδοσιακό κώδικα θεωτολογίας που ισχύει για όλους τους υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε ότι φέτος θα μπορέσουμε να ισχύσουμε ακόμα περισσότερο το κώδικα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πίξτε, μήπως θα θέλατε να πείτε και εσείς δύο λόγια. Ε, ε, Είμαι πολύ σύντομος ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις και εγώ του κυριώτη, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο που συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μου και που είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Μιλήσατε για τη δεοντολογία. το θέμα αυτό δεν νομίζω ότι το έθιξε κανείς μέχρι στιγμής ε, ποτέ Οπότε το θέμα των αντιμαχωμένων συμφερόντων δεν ετέθη κανονικά ποτέ. Νομίζω ότι ο ρόλος ενός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου είναι σαφής, πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και των πολιτών. Και αυτό είναι όλο. Αυτός είναι ο ρόλος μας και σε αυτόν πρέπει να αφιερωθούμε σε ό,τι αφορά τώρα τα προσόντα για την κατάρτιση ε, των ασκούντων τον έλεγχο, ε, θυμάμαι ότι είχα πάρει μέρος ε, πέρυσι στο ελεγκτικό συνέδριο σε ένα διαγωνισμό που αφορούσε, ήταν διαγωνισμός για ελεγκτές χρηματοοικονομικών τομέων και Είχα περάσει πρώτος στον βελγικό διαγωνισμό, ο οποίος τότε είχε ε, επινοηθεί. Τώρα βεβαίως είναι λίγο επαναληπτικός, αλλά στην αρχή ήταν πάρα πολύ αυστηρός και δύσκολος διαγωνισμός. Αυτή τη φήμη είχε. Ε, εν πάση περιπτώσει, έτσι συμβαίνουν τα πράγματα στο Βέλγιο καμιά φορά. Ε, μετά από ένα διάστημα ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να τον βοηθήσω στο γραφείο του και σε μας ε, δεν είναι τα ε, πράγματα ξεχωριστά, δηλαδή τα οικονομικά από την ε, διακυβέρνηση της χώρας, όπως συμβαίνει στη Γαλλία. Στο Βέλγιο είναι στην έθουσα Τρία όλοι οι ελεγκτές συγκεντρώνονται ε, και έχουν ε, ένα κοινό αντικείμενο, ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο εξειδικευμένο αντικείμενο και ασχολούνται με αυτό γιατί, γιατί έτσι γνωρίζονται, μπορούν να συμφάγουν, μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και στη συνέχεια να κρατήσουν μια επαφή για μια πιο αγαστή συνεργασία. Θα θέλατε κάτι να πείτε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. το θέμα είναι το βιογραφικό μου και το από πού προέρχομαι ε, στην συνεργασία μαζί σας. Είδα στο παρελθόν μου αλλά και στην σημερινή μου δουλειά ε, το πιο σημαντικό ήταν η εμπειρία μου και βεβαίως ε, έχει σχέση άμα δείτε το βιογραφικό μου, με τη διαχείριση. Ε, στο management ήταν η κυριότερη απασχόλησή μου τα περισσότερα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια μακρά εμπειρία συνεργασίας με τους εμπειρογνώμονες σε οποιοδήποτε τομέα. Γιατί ε, αν έχει κανείς το ε, management μία κάποια εμπειρία σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να έρχεται σε επαφή με διάφορους εμπειρογνώμονες που αφορούν το δικό του τομέα αλλά και όλους τους άλλους τομείς. Και αυτό είναι ένα σημείο που θέλω να τονίσω. Η δεύτερη εμπειρία που είναι πολύ βοηθητική και θετική για μένα πιστεύω είναι ότι έχω δουλέψει στο δημόσιο τομέα στη Σουηδία. Ε, και επίσης έχω υποστεί επίσης έλεγχο και είναι μια θετική εμπειρία για τον ίδιο τον ελεγκτή να έχει υποστεί έναν έλεγχο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάλα, θέλετε κάτι να πείτε ως συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, τελειώνοντας, περατώνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε όλες τις ερωτήσεις και τα σχέδια και τα σχόλια των ε, διαφόρων συντρόφων μου, ανδρών και γυναικών και πάνω σε αυτά τα τελευταία σχόλια βλέπουμε ότι ο επαγγελματικός χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός και ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου πρέπει να χαρακτηρίζονται από πολυμορφία και από πολλαπλές ε, λειτουργίες ε, δυνατότητες πολλαπλών λειτουργιών ούτως ώστε να έχουν διαφορετικές απόψεις ε, για να μπορέσουμε να ε, έχουμε μια σωστή επιρροή στις κυβερνήσεις, στις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Τώρα η Ευρώπη διανύει μια κρίση και σε σχέση με αυτά που είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ποικιλομορφία απόψεων και να υπάρχει αυτή η θέση διαφορετική των διαφόρων μέλων μέσα στον χώρο των ελεκτικών ευρωπαϊκών, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, είναι λοιπόν εντελώ διαφορετικές ε, οι θέσεις του κυρίου Πίνστεκ από του κυρίου Καλδέρα και των άλλων. Και αυτό ακριβώς παρόλο που η, η κατάρτισή του είναι καθαρά τεκτική, τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε ότι χρειάζεται αυτή η ποικιλομορφία. Θα λάβουμε λοιπόν αντίστοιχα τη σωστή απόφαση. Ευχαριστώ. Ε, έτσι φτάσαμε στο πέρας αυτής της ακρόασης για τα τρία μέλη ε, του συνεδρίου. Διακόπτουμε τώρα τη συνεδρίαση για τρία λεπτά, τέσσερα ας πούμε, λέει ο Προεδρεύων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I reopen Να ξαναξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, λέει ο πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ. Να καλωσορίσω ορίσω τον κύριο Ότμπο, ο οποίος είναι υποψήφιος, ε, τον οποίο προτείνουν οι αρχές της Δανίας. Να προτείνω να μας μιλήσει για πέντε λεπτά και αυτός και μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της εισηγήτριας και μετά θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους βουλευτές. Έχουμε 40 λεπτά. Έχετε το λόγο κύριε Ορμπό. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και μπορείτε να μιλήσετε ό,τι γλώσσα θέλετε. Μου ζήτησαν να μιλήσω αγγλικά, άρα θα μιλήσω αγγλικά εκτός αν μου τεθούν ερωτήσεις στα δανέζικα όπου θα απαντήσω και στα δανέζικα. Χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής εκ νέου ως υποψήφιος για το ελεγκτικό συνέδριο. Έχω παρευρεθεί εδώ σε αρκετές ε, περιστάσεις το 2007 την τελευταία φορά συνοδεύοντας την Δανέζικη Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ προσδοκώ να γίνω μέλος της, ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ολοκλήρωσα τις σπουδέ μου στο Πανεπιστήμιο της ε, Κοπενχάγης. Ξεκίνησα να εργάζομαι στις δανέζικες αρχές ε, εκτός από τέσσερα χρόνια τη δεκαετία του 80 που εργάστηκα για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο από το 1995 Είμαι στο Ελεγκτικό Συνέδριο και χαίρομαι που εργάζομαι με την Πολιτική Επιτροπή γιατί στη Δανία η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών στο Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει ερωτήματα προς το ελεγκτικό στην ελεκτική υπηρεσία και υποχρεώνεται λοιπόν ε, να υποβάλει αναφορές προς την Επιτροπή αυτή. Είναι σημαντικό τμήμα του, της δουλειάς της ελεγκτικής υπηρεσίας οι εξαιρετικέ σχέσει εργασία με, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ε, προσδοκίε της ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία στην ε, καριέρα μου. Θα γνωρίζετε ότι η Δανία συγκαταλέγεται στις χώρες που υποβάλλουν ετήσια γνωμοδότηση για τα ευρωπαϊκά έσοδα και έξοδα και αυτό για χρονική περίοδο 5 ετών. Επειδή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους δανούς και τους δανούς πολιτικούς. Άρα η γνωμοδότησή μας ε, ακολουθεί την ίδια διατύπωση όπως και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ε, δαπανούμε επιπλέον χρηματοδότηση στην Δανία για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η έκθεση αυτή χέρι υψηλού κύρους από την Δανέζικη Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τονίζει τα θέματα αυτά τα οποία χρήζουν βελτίωση στην Δανία. Είμαι πεπισμένος ότι το γεγονός ε, ότι εστιαζόμαστε σε θέματα ευρωπαϊκών εσόδων και εξόδων έχει βελτιώσει την διαχείριση των ε, κονδυλίων αυτών στην Δανία και έχει βελτιώσει την ποιότητα των ελέγχων και έχει βελτιώσει συνολικά τις γενικές δαπάνες και το επίπεδο χρήση των δαπανών αυτών, καθώς και την ε, συλλογή εσόδων στην Δανία. Επίση να υπογραμμίσω ότι ε, μια ελεγκτική υπηρεσία σε κάθε κρατό μέλο θα πρέπει να εργάζεται στενά με του συναδέλφου του ομολόγου από άλλε χώρε. Μπορεί να έχουμε μονοπόλιο στη χώρα μας, αλλά αν θέλουμε να βελτιωθούμε θα πρέπει να συγκρινόμαστε με τους συναδέλφους από άλλε χώρες και χαίρομαι που στην ελεγκτική υπηρεσία της Δανίας αυτό αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Η συνεργασία με, άλλα, με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένη του ελεγκτικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού και τα τελευταία 8 χρόνια θέλουμε, έχουμε αφιερωθεί στην κατάρτιση διεθνών προτύπων για τους δημόσιους ελέγχους μία σειρά α, τέτοιων προ, προδιαγραφών εγκρίθηκαν πέρσι. Αυτό τι σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες παγκοσμίω μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προδιαγραφές και να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντας αυτές τις προδιαγραφές, εφαρμόζοντάς τις, εφαρμόζουν τα σωστά πρότυπα. Είμαι συνηθισμένος στην ανεξαρτησία, στην ανεξάρτητη δράση μου. Το ίδιο πιστεύω ισχύει και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και όπως προείπα, νομίζω ότι αποτελεί βασικό ζήτημα για το ελεγκτικό συνέδριο να βρίσκεται σε άριστες εργασιακές σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, όπως αντίστοιχα γίνεται και με την Εθνική Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην Δανία. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω στην εισαγωγή μου είναι ότι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να λάβω μία θέση στο ελεγκτικό συνέδριο είναι η διεθνής πρόκληση. Η πρόκληση να εργαστώ σε ένα διεθνέ πρόσωπο. Έχω εργαστεί τέσσερα χρόνια ω ε, νεαρό, αν θέλετε, στο Ελληνικό συνέδριο. Ε, μου προκαλεί την ε, περιέργεια και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερη χρονική στιγμή με την κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πιο πολύ. Βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι το ελεγκτικό συνέδριο κινείται προς την ε, κατεύθυνση συνεργασίας με τις εθνικές υπηρεσίες. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί την εξέλιξη την θεμητή. Σας ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρο. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω εν είδη εισαγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τον κύριο Ότμπο για τις πληροφορίες του. Θα ήθελα πάντως να τον ρωτήσω και είναι αλήθεια ότι στο βιογραφικό σας εμφανίζονται κάποια σημεία που αφορούν την εξαρτησία σας σε σχέση με κάποια τεκτενόμενα στη Δανία. Παρ' όλα αυτά όμως, πέρσι συνέβη κάτι σε σχέση με την δική σας ευθύνη ως ε, γενικού ελεκτή. Είχαμε το σκάνδαλο ενός συγκροτήματος οικοδομικού που λέγεται Derbien όπου το Εθνικό Ελεκτικό Συνέδριο αναγνώρισε ότι δεν είχε ελέγξει και δεν είχε ακολουθήσει τις υποχρεωτικές οδηγίες που θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει όσον αφορά τον έλεγχο του κόστους του κτηρίου αυτού που φαίνεται να εκτοξεύτηκε στα ύψη. Έφτασε το 1 δισεκατομμύριο ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το ποσό, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται. Είπατε ότι το Κοινοβούλιο είχε κάνει κάποιο λάθος, όσον αφορά τον έλεγχο δηλαδή, αυτή τη υπόθεση και όπως καταλαβαίνετε αυτό μας ανησυχεί, γιατί ε, είναι αλήθεια ότι η χώρα σας είναι υποδεχματική όσον αφορά κάποιες προποθέσει και όρου που απαιτεί από τι χώρε μέλη επιτροπή μα. Αλλά αυτή η περίπτωση είναι διάζουσα, επειδή εσεί είστε υποψήφιο και το γεγονό ότι πριν από ένα χρόνο θα έπρεπε να είχατε αποδείξει ή να αναγνωρίσετε ότι είχατε διαπράξει ένα σημαντικό σφάλμα όσον αφορά τον έλεγχο ενός οικοδομικού οργανισμού που προκάλεσε προβλήματα στον προπολογισμό. Αυτό βεβαίω μα ανησυχεί. Θα ήθελα λοιπόν να μα δώσετε κάποιες ε, διευκρινήσει. γιατί έλεγαν κάποιοι στον δανεικό τύπο ότι εσείς αναζητούσατε απασχόληση εκτός Εθνικού Ελεκτικού Σώματος ακριβώς για να διαφύγετε από αυτή την υπόθεση τη σκανδαλώδη. Ευχαριστώ πολύ. Αληθεύει ότι μερικά χρόνια πριν η εταιρεία τηλεόρασης της Δανίας ε, ε, κατασκεύασε καινούρια νέα κτίρια και υπήρξε μια υπερβολική δαπάνη σε αυτόν τον τομέα. Είχε χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη ε, στον προϋπολογισμό, αλλά τα το 4% των ε, κτηρίων αυτών ε, εμένα να χρησιμοποιείται και βάσει των διεθνών προδιαγραφών κατατίσαμε μία, ε, έκθεση, με μία έκθεση και είπαμε ότι δεν είχε, είχαν πληρωθεί οι όροι και πρέπει να πούμε ότι μαζί με την... Μαζί το Υπουργείο δράσαμε από κοινού και καταχωρήθηκε αυτή η υπόθεση. You will all know that I was wrong. We all made mistakes. And if ε, ε, υπήρχαν λοιπόν ορισμένα λάθη που κάναμε σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι εντελώ διαφορετική νομίζω αυτή η περίπτωση με το γεγονός ότι τώρα είμαι υποψήφιος για το Ελεγκτικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Καμία σχέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σανγκάτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω δύο ερωτήσεις να σας θέσω. Η πρώτη αφορά τις γραπτές ε, απαντήσεις, τις ερωτήσεις που τέθηκαν σε σχέση με, τις, ε, με τους ελέγχους επιδόσεων. Λέτε ότι όλες οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, στόχους, ε, πρέπει να έχουν στόχους απαραίτητους και επαρκείς, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικός έλεγχος από πλευράς ε, ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό όμως είναι σοβαρό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έλεγχο προσόντων αποτελεσματικότητας να ακολουθήσουμε αυτή την πρότασή σας. Μπορείτε να εμβαθύνετε επ' αυτού, για... σας παρακαλώ. Και το δεύτερο ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι το εξής έχει σχέση με την θέση σας εδώ. Όταν διαβάζει κανείς το βιογραφικό σας διαπιστώνει ότι σε σχέση με άλλους έχετε μια πραγματική παράδοση, δηλαδή στον έλεγχο δουλεύετε εδώ και πολύ καιρό ήσασταν γενικός ελεγκτής ε, στο, του ελεγκτικού συνεδρίου και δεν έχετε καμιά πολιτική σταδιοδρομία από πίσω σας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πήρατε μέρος σε πολιτικές ιστορίες. Έγινε λόγος για τον Ντέμπιν ε, και ε, υπήρξε και υπερπληρωμή των ε, ιδιωτικών νοσοκομείων, των κλινικών. Το κράτος στη Δανία είχε δώσει υπερβολικά πολλά χρήματα σε κλινικές, είχε δαπανίσει πολύ σημαντικά ποσά και ακούστηκαν ισχυρές επικρίσεις επ' αυτού και είχε υποθεί για παράδειγμα ότι χρειαζόταν πολύ χρόνος ώσπου να έρθουν στα χέρια σας τα απαραίτητα έγγραφα και δεν μπορούσατε να ασκήσετε σωστό έλεγχο κτλ το Βρετανικό, ε, το, συγγνώμη, το Δανικό Κοινοβούλιο, το Folketing, είχε παρέμβει τότε τι θα γίνει λοιπόν στη συνέχεια με την παρουσία σας, θέλετε ενίσχυση με την παρουσία σας του Ελεγκτικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ή θέλετε να γίνει, ε, θέλουν να απαλλαγούν από εσά τη Δανία. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Το πρώτο ε, ερώτημα για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, δηλαδή αν χρειάζονται επαρκή και ικανά αποτελέσματα, αν υπάρχουν οι απαραίτητες απαιτήσει για να πάρει ένα σχέδιο βοήθεια. Τι χρειάζεται στο, στη Δανία για μένα, δεν υπάρχουν αρκετές ε, απαιτήσει σε σχέση με τα αποτελέσματα σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε διοικητικό επίπεδο. Δεν λέγεται με μεγάλη σαφήνεια τι είναι οι στόχοι, τι πρέπει να πετύχει κανείς με τα διαθέσιμα ποσά. Και αυτό δεν αφορά μόνο το πολιτικό σκέλος, αλλά και το διοικητικό. Γίνεται θέμα συνέχεια για το input, δηλαδή για την ποσότητα των χρημάτων που θα τεθούν σε διάθεση και σε χρήση. Και δεν μιλάμε ποτέ για τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε, για τους στόχους. Εάν το έχω γράψει αυτό στην απάντηση, τη γραπτή που σας έδωσα. Ε, το έπραξα γιατί έχει κανείς αυτή την εντύπωση όταν ελέγχει τα σχέδια που υποβάλλονται για βοήθεια και από πλευράς Δανίας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θέλει να η αρμόδια αρχή να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στέλνοντάς με εδώ. Δεν θέλει να αποδυναμώσει το Ευρωπαϊκό, ε, συγγνώμη, το Δανικό Κοινοβούλιο. Θέλει να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό στέλνοντάς με εδώ. Ε, όταν κανείς ε, λοιπόν είναι γενικός ελεγκτής ε, ε, της Δανίας σε ένα εθνικό επίπεδο εν πάση περιπτώσει υφίσταται επικρίσεις και από τους υπουργούς και από την κυβέρνησή του. Αυτό είναι σωστό. Ο Υπουργός Υγείας τον οποίο επικρίνατε και επικρίναμε δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την κατάσταση όταν ξέσπασε αυτή η υπόθεση και όταν τελικά περατώθηκε η υποστήριξη πήγε στο ελεγκτικό δανεικό συνέδριο. Ε, αν έχουμε τις σωστές πληροφορίες που πρέπει να έχουμε ως ε, ελεκτικό δανεικό συνέδριο ή ως ευρωπαϊκό ελεκτικό συνέδριο πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε μια εργασία ποιότητας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ πολύ τον Δανό εκπρόσωπο. Θα ήθελα να θέσω μια εντελώς διαφορετική ερώτηση γιατί είναι ο πρώτος εξωτερικός υποψήφιος που ακούμε σήμερα ε, και φέρνει ε, καινούριες φρέσκες ιδέες στην ομάδα των ε, ελεγκτών ποια είναι η εμπειρία που έχετε πέρα από το δανεικό ελεγκτικό συνέδριο ε, και τι αλλαγές θα θέλατε να επιφέρετε, τις πιο σημαντικές στο ελεγκτικό ευρωπαϊκό συνέδριο. Ε, θα είναι πιο πολύ εσωτερικοί ή εξωτερικοί οι παράγοντες ε, αλλαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την πιο στενή συνεργασία με τις εθνικές υπηρεσίες για το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να εξαρτάται από τους εθνικούς ομολόγους προκειμένου το ελεγκτικό συνέδριο να έχει πιο πολλούς πόρους για τα πιο σημαντικά καθήκοντα τα οποία θα ανακύψουν. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Κρίση, κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα έπρεπε και θα χαρώ να δω αυτή την εξέλιξη, να συνεργαστεί πιο στενά με τι εθνικέ ε, υπηρεσίε για να υποβάλει σχετικέ εκθέσει και αναφορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμμετάσχει στι εξέλιξει αυτέ στο μέλλον. Ναι, συμπληρωματική ερώτηση τη κυρία Ιβάνοβα. Μάλιστα, ακούσαμε για τη συνεργασία με τι εθνικέ ελεγκτικέ αρχέ, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Κοκομπού. Τι πιστεύετε για το θέμα αυτό. Απάντηση. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή σας αποτελεί το πιο σημαντικό εταίρο για το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, σημαντική η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ε, μπορώ να φανταστώ οτιδήποτε άλλο παρά εξαιρετικέ ε, σχέσεις εργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι η Επιτροπή σας εδώ, όπως και η αντίστοιχη Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, της Δανίας, χρειάζεται πιο πολλές εκθέσεις, για παράδειγμα για την χρηματοοικονομική κρίση. Και αυτό θεωρώ αποτελεί μείζωνα πρόκληση για την, το ελεκτικό συνέδριο, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε δηλαδή στις ανάγκες της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρέσλε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η κυρία Ιβάνοβα. Θεωρώ και εγώ ότι από αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας ε, έχουμε μια κενή σελίδα και αυτό είναι κρίμα γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ξέρω ότι δεν θα μπορέσετε να μας αποφύγετε. Εγώ είμαι εδώ από το 2004 και έχω δει πάνω από 20 υποψηφίους ε, στο ελεγκτικό συνέδριο και πολλές υποσχέσεις έχουμε ακούσει ότι θα είμαστε καλύτεροι φίλοι, αλλά αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Άρα θέλουμε να υπάρχουν και κάποια τεκμήρια. Μία γενική... Ο γενικός ελεγκτής τι ακριβώς κάνει. Τρίτη ερώτηση. Αυτά που ανέφερε η κυρία Σέντερ σε ό,τι αφορά το θέμα με τα κτίρια, πώς ακριβώς ε, διαμορφώθηκαν, υπήρχαν φωνές που ζήτησαν παρέτηση, επίσης θέματα συγχρηματοδότησης στην Δανία. Ένα παράδειγμα που μας εκνευρίσε όλους. Δεν ξέρω αν θα θυμάστε την ακρόαση με την ε, Επίτροπο Φίσερ το 2008, το Δεκέμβριο είχε γράψει ο βοτανικός ε, τύπος τα θέματα ε, για τον Bornholm και τη σχετική συγχρηματοδότηση που είχε υπάρξει εκεί και πόσο ανόητο ήταν το παράδειγμα αυτό. Το δανεικό κράτος είχε συνδράμει κατά 50%. Τώρα ακούσαμε ότι έγινε μία αίτηση για ανανέωση της ε, χιονοδρομικής πίστας στη Δανία, το οποίο είχε θεωρηθεί ανόητο παράδειγμα μιας και ποτέ δεν χιονίζει εκεί. Τι έχετε να μας σχολιάσετε. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Well, your starting point was more... Ρωτήσατε στην αρχή κάτι πιο συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά την υποχρέωση αναφοράς προς την Επιτροπή. Συμφωνώ και ξέρω ότι αυτό έχει αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για, τους, για τα παλαιά μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά εγώ προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ. και να επανέλθω στο θέμα που ανέφερε η κυρία Σέντερ, θα ήθελα να πω ότι αν ε, έχει κάνει κάποιο λάθος μια ελεγκτική υπηρεσία στην Δανία, αυτό είναι γνωστό σε όλους, το ξέρουν ε, οι βουλευτές, ο τύπος, γιατί δημοσιεύεται. Θεωρώ ότι κάναμε σε 16 χρόνια που είμαι στο, στην ελεκτική υπηρεσία, κάναμε ένα λάθος, ένα μεγάλο λάθος. Γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν ασφαλής η κατασκευή αυτή, επειδή είχε α, δαπανίσει το 84% των κοντιλίων και είχε ολοκληρωθεί κατά 88%. Ωστόσο, ε, εκ των υστέρων αποκινούμε την εταιρεία για να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί στον καινούριο προπολογισμό. Συνεργαστήκαμε λοιπόν. Δεν κρύψαμε τίποτα. Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν στην Δανία. Γιατί όπως είπα ήταν καλό το ότι δημοσιεύτηκε το λάθος της ελεγκτικής ε, ε, υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά την χειροδρομική πίστα και το lift δεν γνωρίζω ακριβώς τις λεπτομέλειες. Τώρα κοιτάξτε, στο Bornholm, σε ένα μικρό νησί στην Βαλτική, να δημιουργηθεί ένα lift χιονοδρομικής πίστας όπου δεν χιονίζει, είναι τρελό. Από την άλλη, ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται και τεχνητό χιόνι, αλλά όπως σας είπα δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο έργο, οπότε δεν μπορώ να αποφανθώ. Ingeborg, you να ξαναπάρεις το λόγο. Ναι, είχα ρωτήσει κατά πόσον υπάρχουν, ε, κατά πόσον είχαν ακουστεί φωνές που είχαν ζητήσει να παραιτηθείτε στην Δανία. Όχι. Τίποτα τέτοιο δεν είχε ακουστεί. Νομίζω ότι το να παραδεχτούμε ένα σφάλμα σε 16 χρόνια, όπως είπα και στον κύριο Ζόντεργκαρτ, δεν έχω την εντύπωση ότι θέλει κανείς να με ξεφορτωθεί στη Δανία. Δεν ξέρω αν είμαι αφελής, αλλά πιστεύω ότι το Δανικό Κοινοβούλιο με πρότεινε ω υποψήφιο για να ενισχύσει το ελεκτικό συνέδριο και όχι επειδή θέλουν να φύγω. Thank Ευχαριστώ. Κανείς άλλος βουλευτής που θέλει να θέσει ερώτηση προς τον κύριο Ό,τι πω, θα πάρετε το λόγο στο τέλο κυρία Σέντερ. Δεν, θα, ξέρω, θέλει κανεί άλλο το λόγο. Μάλιστα, ωραία, το λόγο στην συγκεκριά. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεπλάγει να οφείλω να ομολογήσω. Επειδή το γεγονό ότι ο τύπο, αναφέρει ότι έγιναν κάποια σοβαρά λάθη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και ευθύνε. Εμείς κύριε Μπόκη καταλαβαίνετε ότι σας εξετάζουμε εδώ ως μέλος του ελεκτικού, Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Κάποια ευθύνη θα έχετε κι εσείς. Εξάλλου αυτό το αναγνωρίσατε ενώπιον του Δανικού Κοινοβουλίου. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, με ποιο τρόπο, εκτό από τη διαφάνεια στην επικοινωνία, κάτι το οποίο βεβαίως θα χοροπήσει όλους τους πολίτες κλπ. Αλλά κάποια ευθύνη πρέπει να έχει κάποιο και να την αναλάβει τέλο πάντων. Ποιο την, την ανέλαβε. εσεί αναγνωρίσατε ότι ήσασταν ο υπεύθυνο εσεί, ότι ε, κάνετε λάθο, ότι κάνετε λάθο, ε, σοβαρό λάθο, μείζον λάθο. Οπότε διαρωτώ με, εντάξει, να είμαστε διαφανεί, αλλά εκτό από διαφανεί, κάποιο πρέπει να λάβει την ευθύνη του, έτσι δεν είναι. Διαφορετικά τι να πω, εσεί πριν από ένα χρόνο κάνατε ένα μείζον λάθο στη Δανία με ένα κτίριο, αναγνωρίζοντα ότι δεν εφαρμόσατε υποχρεωτικού κανόνε στι υπηρεσίε σα. Το λέει εδώ ξεκάθαρα. Και το, λέτε, και το παραδείξετε κι εσείς εδώ δημοσίω. Και θα σας ορίσουμε εμεί τώρα για να μπείτε ως νέο μέλος στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Καταλαβαίνω ότι η ιδανική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά εμεί, όπω καταλαβαίνετε εδώ, εξετάζουμε το τι θα προσκομίσετε εσεί στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Γιατί μα ανησυχεί το ποιο θα αναλάβει την ευθύνη. Εκτό από την δημόσια αναγνώριση και παροδοχή του μεγάλου λάθου. Εκτό από αυτό, κάποιο θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Αυτό πρέπει να γίνει. Διαφορετικά, εκτιθέμεθα σε περίπτωση όπου εσεί του χρόνου επαναλάβετε το ίδιο σοβαρό μείζον σφάλμα στα πλαίσια του δημοσίου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έγινε λοιπόν αυτό πριν από ένα χρόνο. Δεν βλέπω να αναλαμβάνετε να λαμβάνετε εσείς την ευθύνη και με ένα χρόνο αργότερα ζητάτε να γίνετε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου και μπορεί σε ένα χρόνο εσείς να μας πείτε εντάξει λυπάμαι κάνα πάλι το ίδιο μεγάλο λάθος. Εσείς την ευθύνη σας πώς θα την αναλάβετε. Well, I full responsibility. Εγώ ανέλαβα πλήρη ευθύνη. Ανέλαβα πλήρη ευθύνη για την συγκεκριμένη υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2006, όχι πέρσι. Η υπόθεση αυτή που αναφέρεται αναφέρεται στον έλεγχο της επιχείρησης του 2006. Και όταν μιλήσαμε όταν κάναμε μάλλον την αναφορά μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του, του Δανικού Ελεκτικού Συνεδρίου, θεωρήσαμε ότι η υπόθεση πήγαινε καλά. Εκεί κάναμε λάθος. Και δημοσίως αναγνώρισα ότι η διατύπωση μας ήταν λάθος και θεωρούσαμε ότι δεν έκανα υπέρβαση του προπολογισμού. Οπότε λοιπόν το λάθος αυτό, το σοβαρό λάθος όπως το ονομάσατε, Το αποδέχτηκα και ανέλαβα πλήρη ευθύνη. Και ξαναλέω, ανάγεται στο 2006 η υπόθεση αυτή, όχι στο 2010. Και δεν υπάρχει βολή για το ποιο ήταν υπεύθυνο. Εγώ ήμουν υπεύθυνο και έχω αναλάβει πλήρη ευθύνη. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Θέλετε πάλι το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Να πω ότι ναι, είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε το 2006 αυτή η υπόθεση, όμως στις περικοπές που χρειάστηκε να γίνουν όσον αφορά τη δημόσια τηλεόραση, όσον αφορά εκπομπές κτλ. Εκτός μικροφώνου, η κυρία Γελά. Α, 300 300 εκατομμύρια κορώνες κάθε χρόνο μέχρι το 2010. Το πράγμα λοιπόν είναι επίκαιρο, όχι μόνο επειδή ξεκίνησε το 2006, αλλά επειδή αυτές οι περικοπές οι οποίες έγιναν λόγω ακριβώς του σφάλματος οδήγησε μέχρι, μέχρι το σήμερα. Οπότε, Πρόεδρε, αυτό ήθελα να πω. Να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά τα στοιχεία. Εγώ πάντως δεν θεωρώ σαφές το ότι η αναγνώριση του σφάλματος θεωρείται επαρκής ως ανάληψη ευθύνη τη στιγμή που έχουμε ένα τόσο σοβαρό λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Yes. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω θα πρέπει να θυμάστε ότι εγώ δεν ήμουν αρμόδιος υπεύθυνο για την οικοδόμηση αυτού του κτηρίου. Ήμουν ο ελεκτής. Ανέλαβα πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ελεκτική εργασία. Η διατύπωση ενδεχομένω να σας κάνει να πιστεύετε ότι ήμουν υπεύθυνο για την οικοδόμηση του κτηρίου. Ναι, ναι, βεβαίω, για, για τον έλεγχο. Ναι, ναι, για τον έλεγχο Βεβαίω, για τον ελεγχό είχαμε εφαρμόσει διεθνεί προδιαγραφέ καθ' όλη τη διαδικασία. Αλλά η διατύπωση αφορά ένα σφάλμα μια συγκεκριμένη χρονιά όπου θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχαν υπερβάσει στον προπολογισμό. Είπα λοιπόν ότι και παραδέχτηκα ότι ο προπολογισμό εφαρμοζόταν και αρκούσε για την ολοκλήρωση της οικοδόμησης. Αλλά δεν ήταν έτσι. Η υπεύθυνη για την υπέρβαση του προπολογισμού δεν ήταν οι ελεκτέ. Ευχαριστώ. Μήπω κάποιο άλλο επιθυμεί το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Τότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κάνουμε ένα διάλειμμα για λίγα λεπτά. τόρτο. θες mm.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 Could I ask everybody to resume their seats? Αν θέλετε καθίστε λίγο. Μπορείτε να καθίσετε. I τη συνεδρίαση και χαιρετίζω τον κύριο Γουάν Φρανσίσκο Κορώνα Ραμόν ο οποίος έχει οριστεί από την Ισπανική κυβέρνηση ε, ως μέλος ε, ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Δίνουμε λοιπόν πρώτα τον λόγο στον υποψήφιο για πέντε λεπτά, ούτω ώστε να μας εξηγήσει τις προθέσεις του ως μέλος του, στο Λουξεμβούργο του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια του χρόνου που έχω θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα Εγώ είμαι ένα τεχνοκράτης. Εργάστηκα σε θέματα ελέγχου και δημοσίων οικονομικών. Ιδιαίτερα από το που τέλειωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο ξεκίνησα τη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης στο τμήμα των Δημοσίων Οικονομικών και στη συνέχεια μέσω διαγωνισμών. Ανέβηκα βαθμίδες μέχρι το 1993 όπου έφτασα στο μέγιστο βαθμό σύμφωνα με τον Ισπανικό κανονισμό που είναι τακτικός καθηγητής Μοσίων Οικονομικών. Εργάστηκα σε διάφορα πανεπιστημία τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά στην Βαρκελόνη, στις Βαλεαρίδες και μάλιστα κάποια εποχή και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και με μεγάλο τμήμα της δραστηριότητά μου ε, αφορούσε την ε, διδασκαλία και την έρευνα στα δημόσια οικονομικά. Συμμετείχα σε διάφορα διεθνή προγράμματα, ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική με την Νοτιοαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και συμμετείχα σε συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούσαν συγκεκριμένες χώρες δηλαδή και κυβερνήσεις που μέσω λόγω ακριβώ αναγνώριση του προσωπό μου ανέθεσαν διάφορες εργασίες. Όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών, άρχισα να δουλεύω ω ελεκτής αμέσω μετά την αποφύτησή μου. Ήμουν στο Grand ω junior ελεκτής για δύο χρόνια. Μετά έγινα ελεκτής senior και αυτό μου επέτρεψε να είμαι ένας από τους ιδρυτές του επίσημου Μητρώου Ελεκτών που απετέλεσε τον πρώτο επίσημο οργανισμό που δημιουργήθηκε στην Ισπανία για την ρύθμιση και προάσπιση του επαγγέλματος του ελεκτή. Στη συνέχεια ήμουν ένας από τους δημιουργούς του Μητρώου Οικονομολόγων Ελεκτών και το οποίο είναι ένα όργανο το οποίο σχετίζεται με το Σωματείο Οικονομολόγων, το Σώμα Οικονομολόγων της Ισπανίας. Στη συνέχεια είχα αναλάβει διάφορες εργασίες στα πλαίσια του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών και παραδειγματικά να σας πω ότι κάποια χρόνια ήμουν στο Διοικό Συμβούλιο του Ισπανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Αναλυτών και ήμουν εκπρόσωπος του επαγγελματικού κλάδου των ελεκτών όσον αφορά τους οικονομικούς αναλυτές. Βλέπετε λοιπόν κατά συνέπεια ότι το προφίλ μου το επαγγελματικό είναι τεχνοκρατικό και να πω επίσης ότι κατά διάρκεια εκείνης περίοδου συνεργάστηκα συχνά με την Ισπανική κυβέρνηση κατά διάρκεια διαφόρων κοινοβουλευτικών θητιών και αφού είμαι και καταναλωνός συνεργάστηκα τακτικά με την τοπική καταναλωτική κυβέρνηση την Generalitat de Catalunya. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε και ελπίζω στο μέλλον να είμαι σε θέση να διτελέσω ένα πολύ καλό έργο να επιτελέσω ένα πολύ καλό έργο στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο κάτι το οποίο για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία ως εμπειρογνώμονα των δημοσίων οικονομικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει και ο Πρόεδρος ο λόγος στην εισηγήτρια την κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κορώνα Ραμόν για αυτή την παρουσίασή του. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ένα προφίλ το οποίο με εξέπληξε γιατί είναι καθαρά επαγγελματικό που έχετε ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασία με πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Έχετε μια θαυμάσια διαδρομία Και βλέπω ότι στο βιογραφικό σας ότι είστε μέλος και του καταλανικού τμήματος της, του Ιδρύματος ΦΑΕΣ, στο οποίο προεδρεύει ο κύριος Αθνάρ. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσετε κάπως τον ρόλο σας και τη συμμετοχή σας σε αυτό το Ίδρυμα. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία σας με την τοπική καταναλωτική κυβέρνηση, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο εσείς θα ήσασταν διατεθειμένους, γιατί αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου θα εργαστούμε μελλοντικά, να συνεισφέρετε σε περίπτωση που οριστείτε ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου στην προσέγγιση της εξαγωγής οικονομικού ελέγχου με τις τοπικές κυβερνήσεις όπου λόγω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να ελέγχονται και τα κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία. Νομίζω ότι ένα τομέα αυτό που θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου και να πω επίση, να πω μάλλον πάλι ότι είναι εντυπωσιακό το βιογραφικό σας, η σταδιοδρομία σας, η τεχνοκρατική. Και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία σας η περιφερειακή θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το συνέδριο. Θα ήθελα να τα διευκρινίσετε λοιπόν αυτά. Ναι, λέει ο πρόεδρο, έχετε το λόγο. Ναι, βεβαίω, λέει ο κύριο Κορονάραμον, για το πρώτο σημείο που θίξατε. Οι πληροφορίε που έχετε είναι σωστέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βάζω συνήθω αυτό στο βιογραφικό μου, για αυτό το ίδρυμα που αναφέρατε, γιατί δεν έχει οικονομική άλλη δραστηριότητα. Και πράγματι η παρουσία μου ως μέλος σε αυτό το Ίδρυμα οφείλεται στο ότι Ο Ζωζέ Πικέ ήταν υπουργός εξωτερικών και υπουργός οικονομικών στην, ε, στην Ισπανία. Ο Ζωζέ Πικέ ήταν φίλος προσωπικός ε, από την Βαρκελόνη και πρόεδρος του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος στην Καταλωνία. Ως προσωπικός λοιπόν φίλος μου ζήτησε να γίνω μέλος αυτού το Ίδρυμα, κάτι το οποίο αποδέχτηκα και βεβαίως να καταστήσω σαφές ότι δεν είχα καμία πολιτική σύνδεση ε, με το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα γιατί ανέκαθεν προσπαθούσα να συνεργαστώ με όλα τα ισπανικά πολιτικά κόμματα που μου το ζήτησαν. Αποδέχτηκα λοιπόν την πρόσκλησή του για συμμετοχή στο Ίδρυμα αυτό και θα αποδεχόμουν να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα που είχε αυτά τα χαριστικά και που προχώταν οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που ρωτούσατε για την ε, καταλανική κυβέρνηση, γιατί πραγματικά ε, γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα που αφορούν και την τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας αλλά και την αντιπολίτευση και η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενόχλησα ή παρενόχλησα τις κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργάστηκα και αυτό το έχει αναφέρει και ο τοπικός τύπος. Γιατί πάντοτε αναζητούσα την μέγιστη αποτελεσματικότητα και μέγιστη αποδοτικότητα τη οικονομία όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, κατά το οποίο χρηματοδοτούμε όλοι μας. Κατά συνέπεια, δεν έχω καμία αντίρρηση, αν χρειάζεται ή αν χρειαστεί, να δράσω με τελείω ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο στα πλαίσια τη ασκή οποιοδήποτε ελέγχου είτε πρόκειται για εθνική είτε πρόκειται για περιφερειακή κυβέρνηση. Να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι λόγω ακριβώς της τωρινής περίπλοκης δομής της Ένωσης και των χωρών της Ένωσης η ενίσχυση του ελέγχου και των σχέσεων με τα λεκτικά συνέδρια και τα κρατικά ή και τα υποκρατικά όπως στην περίπτωση της Ισπανίας οι αυτόνομες περιφερειακές δηλαδή δομές ελεκτικών συνεδρίων αυτό νομίζω είναι απόλυτα απαραίτητο ώστε η δουλειά του ελεκτικού συνεδρίου να είναι χρήσιμη και να βοηθά το Κοινοβούλιο να ασκεί τον απαραίτητο νομικό και πολιτικό έλεγχο. Οκ, okay, okay, λέει ο Πρόεδρος. To Τώρα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές και ε, καταρχάς την Ingeborg Γκρέσλε. Ευχαριστώ καθηγητή Ραμόν. Δεν κατάλαβα από τα έγγραφα ποια είναι η επαγγελματική σας δραστηριότητα, η τρέχουσα επαγγελματική σας δραστηριότητα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω πιο πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Επίσης είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Πριν από τρεις ημέρες έγιναν εκλογές στην Ισπανία και η σοσιαλιστική κυβέρνηση ιτήθηκε η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις συνθήκες φυσικά, έχει ε, την ευθύνη να θερήσει τον υποψήφιο, αλλά το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα αυτό στην νέα ε, κυβέρνηση. Στην ομάδα μου επέμεινα ότι η υποψηφιότητα αυτή δεν μπορεί να ισχύει για υποψηφίους που έχουν ε, δεν ξέρουμε δηλαδή κατά να έχει το, η παλιά κυβέρνηση το δικαίωμα να υποβάλει υποψήφιο. Τρεις ημέρες όμως μετά, την, ε, μετά τις εκλογές θέλω να δώσω στη νέα κυβέρνηση την δυνατότητα να υποβάλει τον νέο υποψήφιο. Ποιος σας ε, διόρισε ως υποψήφιο λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει και θα θέλω να καλέσω τους ε, συναδέλφους να δώσουν το δικαίωμα στη νέα κυβέρνηση να υποβάλει τον υποψήφιο, γιατί έχει αναλάβει τα καθηκοντά της εδώ και τρεις ημέρες. Υπάρχουν καλοί λόγοι να μας ε, οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να περιμένουμε με τον διορισμό σας. Ε, επίσης, να σας ρωτήσω πώς φαντάζεστε τις σχέσεις σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο στο Λουξεμβούργο, απέχει κάπως από τις Βρυξέλλες. Αν δεν υπάρχει προσπάθεια λοιπόν για τις επαφές με το Κοινοβούλιο, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Πώς ε, έχετε εργαστεί και συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλετε να απαντήσετε κατευθείαν, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα, ωραία. Ναι, σε σχέση με την τωρινή μου επαγγελματική ιδιότητα, αυτή είναι διητή Αφενός εργάζομαι ως τεχνικός διευθυντής σε έναν οργανισμό που ονομάζεται Ιστιτούτο Επαγγελματικής Επιχειρηματικότητας ένας οργανισμός δηλαδή των πιο σημαντικών οικογενειακών ε, επιχειρήσεων που, υπάρχει, που υπάρχουν στην Ισπανία και που ασχολείται με την παροχή συμβουλών σε τεχνικό επίπεδο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εργάζομαι εκεί part-time. Όπως και σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, όπου διδάσκω το μάθημα των δημοσίων οικονομικών. Στο τμήμα δικαίου, πολιτικής επιστήμης και οικονομικών όπως επίσης διδάσκω και στο δακτορικό αυτού του πανεπιστημίου. πανεπιστημίου. Για το τεχνικό κομμάτι της δραστηριότητά μου, όπως αναφέρεται στο βιογραφικό, είναι προφανές ότι εγώ δεν βρίσκομαι εδώ επειδή ανήκα ή ανήκω σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Είμαι εδώ καθαρά χάρη στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και στον τομέα του ελέγχου όπως και στον τομέα των δημοσίων οικονομικών. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που από το 1984 συνεργάστηκα μετά από ετοιμά με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από την Ισπανία, την Σοσιαλιστική του Φελίπε Γκονθάλεθ, την, της, του Λαϊκού Κόμματος Αθνάρ και μετά το Σοσιαλιστικό σοσιαλιστική κυβέρνηση του Θαπατέρο και στην Καταλωνία ακριβώς το ίδιο. Συνεργάστηκα με όλε τις κυβερνήσεις που πέρασαν από την Καταλωνία από το 1984. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν με κάλεσαν να συνεργαστώ μαζί τους για πολιτικούς λόγους, αλλά χάρη στο βιογραφικό μου και στις προδιαγραφές που και σε απαιτήσει που θέτηκε με συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Όσον αφορά τώρα τι νομικέ δραστηριότητε, υπάρχουν κάποιε διαδικασίε με κάποια χρονοδιαγράμματα και προθεσμίε που εγώ βεβαίω δεν είμαι το καλύτερο άτομο να σα αναφέρω, αλλά που θεωρώ ότι τηρούνται βλαβικά και είναι αλήθεια ότι είχαμε εκλογέ, αλλά η τωρινή Ισπανική κυβέρνηση μέχρι να συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις κάλπες πριν από τέσσερα χρόνια και η διαδικασία επίσης λειτουργίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά διάρκεια της θητείας μιας ε, κυβέρνησης, τότε προφανώς απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι η Υπουργός Οικονομίας και πρώτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αυτά που κάνει είναι σύμφωνα με την νομιμότητα. Για το τρίτο ερώτημα, είναι ενδιαφέρον οι σχέσει δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μια προσωπική άποψη επ' αυτού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ στενές, καταβάλλονται σαφώ προσπάθειες, αλλά ίσω να μην αρκούν. Γιατί σε τελική ανάλυση ένα τεχνικό όργανο το ελεκτικό συνέδριο που αυτό που κάνει δεν είναι τίποτα άλλο από το να προσφέρει πληροφορίε και χρήσιμες αξιολογήσεις ώστε να ασκήσει κατάλληλα τη δραστηριότητα το Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόσταση μεταξύ Βρυξελό και Λουξεμβούργου ε, που δεν είναι θα πρέπει να αποτελεί ένα μειονέκτημα. Αντίθετα θα πρέπει να ενισχύσουμε στο μέγιστο τη σχέση αυτή μέσω των εισηγητών και όλων των εμπλεκομένων. Πάντω, εγώ ω μέλο του συνεδρίου θα είμαι πάντοτε στην διάθεση των μελών του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα στην διάθεση της δικής σας επιτροπής της Κοκομπού. Uh, ε, is it a point of order or is it... Διαδικαστικό, κυρία Σέντερ. No, okay. In that case, I give the... Αν όχι, θα δώσω το λόγο και πάλι στην, θα στην κυρία Γκουτιέρες Κορτινά. Muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα προσόντα του κυρίου Κορώνα όπως και άλλων που θα μπορούσαν να ήταν υποψήφοι, είναι προσόντα μια ακαδημαϊκής καριέρας. Όμως εγώ να αναφέρω την ανησυχία μου και δεν έχω αφιβολίε για την επαγγελματική σας ικανότητα, αλλά θα ήθελα να θίξω τα εξή. Θα ήθελα να αναβάλουμε αυτόν τον διορισμό μέχρι να υπάρχει συνένεση και να ακούσουμε την άποψη της ισπανικής κυβέρνησης που ανέκυψε από τις κάλπες πριν από τρεις μέρες. Νομίζω ότι Έχω εδώ την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης όπου αναφέρεται η πάυση του Θαπατρός Πρωθυπουργού. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε δύο διαφορετικά κριτήρια εδώ που είναι πολύ σημαντικά από τη δημοκρατική σκοπιά. Το ένα είναι νομιμότητα και το άλλο είναι η θεμητότητα. Έχουμε την δημοκρατική νομιμότητα και την δημοκρατική θεμητότητα. Διαφορετική έννοια αυτή. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη, παρόλο που η προηγούμενη κυβέρνηση θα μπορούσε κάτι να συμφωνήσει με την τωρινή και να επιλεχθεί ο κυρίως Κορώνα, δεν έχω αντίρρηση, αλλά θα πρέπει το νόμιμο και το θεμητό να συμβαδίζουν. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ καλό για την προσθέμενη αξία της δημοκρατίας. Και να πω κάτι στον κύριο Κορώνα, το οποίο πράγματι με ανησυχεί. Εδώ δεν υπήρξε συνένεση. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήσασταν στην ΦΑΕΣ, στην Καταλωνία, θα μπορούσε κανείς και το γεγονός ότι θα μπορούσε κανεί να έχει και την σύμφωνη γνώμη τη προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό με και ένα ανησυχώ για το κατά πόσο αδιάκριτα έχει την υποστήριξη όλων ο υποψήφιο. Δηλαδή έχουμε εδώ την υποστήριξη από κάτω το οποίο είναι εκτός κοινοβουλίου. Ένας εκπρόσωπος μιας χώρας θα πρέπει να διακρίνει ξεκάθαρα μεταξύ των πράξεων μιας κυβέρνησης και των πράξεων ή αποφάσεων ή δράσεων ενός ιδρύματος όπως αυτή η ΦΑΕΣ η οποία βεβαίως ε, πρόσκειται στο Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Αυτό μου ανησυχεί λοιπόν. Επιμένω λοιπόν ώστε να αναβληθεί αυτή η διαδικασία, ώστε να έχουμε την απαραίτητη επίσημη συνένεση, γιατί η συνένεση δεν είναι κάτι το μιλταίο, και εξάλλου αυτό θα οδηγήσει τον κύριο Κορώνα να σε θέση να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντά του σε περίπτωση που επιλεγεί από εμά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να σχολιάσετε τώρα αμέσω. Πρόεδρε, να διευκρινίσω κάτι. Απαντώντα αυτό που είπε η κυρία Κορτίνη στο τέλο, να διευκρινίσω ότι θεωρώ ότι ο υποψήφιος δεν έχει μπερδέψει τίποτα. Έχουμε μια πρόταση συνενετική από την κυβέρνηση της Ισπανίας και το γεγονό ότι είναι μέλος στο Ίδρυμα ΦΑΕΣ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έθεσα εγώ, όχι ο υποψήφιο. Να μην υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία. Εγώ ίδιος εξεπλάγιν τα πληροφορίε όπω κάνω για όλου του υποψηφίου και επειδή είδα ότι υπήρχε πρόταση από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο υποψήφιο και επειδή είχαμε μια πολύ καλή τεχνοκρατική ε, σταδιοδρομία, ε, ανέφερα αυτό το σημείο το οποίο με ξέπληξε κάπω. Το διευκρινίζω λοιπόν ότι εγώ ήμουν αυτό που έθεσε αυτό το θέμα και όχι υποψήφιο. Eh, Απάντηση, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο ναι, για το πρώτο τμήμα της ερώτησης ήδη απάντησα, μάλλον απαντήθηκε, και για το δεύτερο τμήμα της ερώτησης εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Η νομιμότητα βεβαίως για ένα βουλευτικό σώμα είναι αυτό που προέχει. Μιλάμε για ένα ελεκτικό συνέδριο που έχει για ένα σώμα μάλλον, συγγνώμη, που έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και δεν έχει πολιτικό προφίλ. Και το γεγονό ότι κατά διάρκεια της ε, σταδιαδρομία μου δεν είχα διασυνδέσεις ε, πολιτικές, νομίζω ότι αυτό από μόνο του εντείνει το χαρακτήρα της ε, σωστή υποψηφιότητά μου για το Ευρωπαϊκό Λεπτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ να απευθυνθώ και, στους προς, και προς τους συναδέλφους ε, όταν ε, εξετάζουμε θέματα του πώς αξιολογούμε την ακρόαση. Γιατί κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Να το επαναλάβω, ίσως. Παρακαλώ να επανέλθουμε στην ακρόαση, να θέσουμε ερωτήσεις στους υποψηφίους και να αποφασίσουμε πώς θα αξιολογήσουμε τελικά τα αποτελέσματα. Να μιλήσω και να θέσω το ερώτημα ίσως για την Ιντανέζικη κυβέρνηση. Αλλά να θέσω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Κόρονα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Προσπαθούμε να μειώσουμε το περιθώριο σφάλματος ε, που διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά την δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ισπανία στο σημείο αυτό πάντα αποτελεί πηγή ανησυχιών. Και ακούγοντα τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό έχει να κάνει κυρίω με την διοικητική δομή στην Ισπανία. η οποία συνεπάγεται ότι η διαχείριση των πόρων εναπόκειται σε τοπικό επίπεδο, σε κάποιες περιπτώσεις σε κεντρικό εθνικό επίπεδο, σε κάποιες άλλες και έτσι υπάρχει πρόβλημα κατανομής αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Στις εργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού η Ισπανία αποτελεί ένα σημείο όπου θα πρέπει να εργαστούμε πιο εντελεχώς. Πόσο ανεξάρτητα λοιπόν ε, μπορείτε να αφιερωθείτε στο έργο αυτό, πόσο ανεξάρτητα σε σχέση με τις εθνικές ισπανικές αρχές. Ε, muy bien, muchas gracias. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Τραμών. Συμφωνώ μαζί σας. Ξέρουμε ότι η Ισπανία λαμβάνει πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στο να υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που περιλαμβάνουν περισσότερα σφάλματα από ό,τι συνήθως. Αλλά ως μέλος της Επιτροπής εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν το ποσοστό σφάλματος στην εφαρμογή των στη χρήση των κονδυλίων είναι υψηλό θεωρώ απαραίτητο στο μέτρο του δυνατού να εμβαθύνουμε στη σχέση αυτή μέσω και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης μέσω και των αυτόνομων των Περιφερειακών Ελεκτικών Συνεδρίων τη Ισπανία. Εγώ βέβαια είμαι διατεθειμένο να το κάνω αυτό, όπως οτιδήποτε άλλο βοηθάει τον στόχο μα, ο οποίο είναι η σωστή εκτέλεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Οτιδήποτε θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να το κάνουμε. Ωραία. Κυρία Γιάλα, Σα έχω στον κατάλογο των ομιλητών. Έχετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ επιθυμούσα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση να σχολιάσω αυτό που είπε η προελίσσασα ε, συνάδελφος. Α, μήπως θέλει εσύ το λόγο. Έχετε ερωτήσει ακόμα. Α, ωραία, αφού έχετε ερωτήσεις Έχετε ερώτηση ή όχι, ρωτάει ο πρόεδρο. Είμαστε στα συμπεράσματα. Όχι, όχι, είμαστε ακόμα στο πλαίσιο των ερωτήσεων προ του υποψηφίου. Η κυρία έχει το λόγο. Ο κύριο Ρωτή, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Κορώνα και η ανακοίνωσή του δείχνει ότι είναι εξαιρετική διαδικασία και κατά την άποψή μου πληρεί τις προϋποθέσεις ε, ε, του άρθρου, δηλαδή ε, που μας απασχολεί, των εμπειριών, δηλαδή στον έλεγχο. Εγώ είμαι εισηγητή εξ ονόματο της ομάδας μου. Υπάρχει όμω ένα πρόβλημα νομότυπου χαρακτήρα πολιτικού. νομίζω ότι στην παρέμβασή σα θα ήταν σωστό να εξηγήσετε τις προθεσμίες που έχουμε να με τις οποίες έχουμε να συμμορφωθούμε και είναι θέμα ευθυνών δικό μας. Υπάρχει το δικό σας πρόβλημα που δεν είναι δικό μας και συγγνώμη που σας το λέω αλλά ήταν εκτός θέματος η παρέμβασή σας ως επ' αυτού του θέματος. Νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία. Ο καθένας διαποδίδει άλλες ε, διαστάσεις στον εαυτό του. Ο κύριος Κορώνα έχει μια προσωπικότητα, μια πολύ καλή υποψηφιότητα. Αλλά δεν θέλουν να υπάρχουν παράπλευρες βλάβες μιας πολιτικής ε, φιλονικίας η οποία δεν θα έκανε καλό σε κανέναν. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κανόνες. Εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε το δίκαιο και να μην το σεβόμαστε. Είμαστε πολιτικοί, πρέπει να ασκούμε πολιτική γιατί αυτό είναι το καθήκον μας έναντι των συμπολιτών μας και Έχουμε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος, πολιτικές πληροφορίες. Έγινε και αλλαγή κυβέρνησης ε, στο κράτος μέλος που προτείνει αυτή την εξαιρετική υποψηφιότητα. Ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι συνθήκη, αλλά ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει ότι εάν υπάρχει αντίθεση 40 βουλευτών ε, της αρμόδιας επιτροπής μιας πολιτικής ομάδας, είναι κυρίαρχο το Κοινοβούλιο να αναβάλει την ε, τον ε, διορισμό. Η αλλαγή λοιπόν της κυβέρνησης είναι ένας αποχρόν λόγος, ένα αποχρόν στοιχείο, κενό στοιχείο αποχρόν ούτως ώστε μία από αυτές τις τρεις πολιτικές αρχές, δι, δηλαδή είτε πολιτική ομάδα είτε η Επιτροπή σας, αλλά δεν ξέρω με ποιες συνθήκες θα έπρεπε η Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε να ψηφίσει και να προτείνει στο Κοινοβούλιο να αναβάλει αυτήν την ε, διαδικασία διορισμού, να επιληφθεί το Κοινοβούλιο του θέματος και να μπορούμε να πούμε εάν είναι επαρκή τα στοιχεία που έχουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα κυβερνήσουν την Ισπανία σας ρωτώ, ε, αν έρθουν στην εξουσία θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας. Είναι σαφές το ερώτημα και θέλω να τονίσω ότι θα μιλήσουμε για διαδικασίες και για ποιότητα των υποψηφίων το απόγευμα. Αυτό είναι μια... Σήμερα το πρωί έχουμε την ε, συνεδρίαση που αφορά την πληροφόρηση ε, των... της Επιτροπής μας για την ποιότητα των υποψηφιωτήτων και των υποψηφίων. Θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε παρουσίαση σχετικά με τις απόψεις σας τα υπόλοιπα το απόγευμα. Κυρία Κρέσλε, η Ισπανία εδώ και 10 έτη είναι στην κορυφή όλων των ατασταλιών σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά ταμεία. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και πραγματικά έχουμε μείνει άφωνοι. Το ελεκτικό συνέδριο ως τώρα δεν έχει συνδράμει στην εξέβρεση λύσεως. Γιατί αρνείται να προβεί σε κατονομασία των ε, υπευθύνων, στο naming and shaming. Η Ελλάδα και η Ισπανία ευθύνονταν για το 95% όλων των ατασταλιών. Και τώρα έχει πάρει την θέση της Ελλάδας η Τσεχία. Αυτές οι πληροφορίες όμως είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα αν το, Ισπανικ, το μέλος από την Ισπανία, δεν θυμάμαι το όνομα του απερχόμενου μέλους, αλλά αν το μελλοντικό μέλος από την Ισπανία φρόντιζε να αντιμετωπίσει το θέμα με την ίδια του τη χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να να θίξουμε τέτοια θέματα προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς. Σαφής η ερώτηση λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Αυτό ήδη το κάνω. Όχι μόνο με την τωρινή, αλλά και παλαιότερες κυβερνήσεις ήλθαν σε επαφή μαζί μου και μου ζήτησαν να συνεργαστούμε. Εγώ ακολουθώ κάποιες αξίες ιερές και το γεγονό ότι είμαι Ισπανό επουδενή δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε μου άποψη. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός μου θα προσπαθήσω βεβαίω να δράσω όχι μόνο για το καλό τη Ισπανία, αλλά για το καλό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Ευχαριστώ πολύ. Στα πλαίσια των ερωτήσεων, να πω το εξή. Με τι δυσκολίε που θα έχει ένα ελεκτή με την Ισπανική κυβέρνηση και με τι περιφέρειες κάτι το οποίο από μόνο το υπαρκεί για να γίνει περίπλοκη εξολόγηση του ελέγχου των ισπανικών δαπανών. Δεν πιστεύετε εσείς ότι θα έχει περισσότερη δύναμη η δουλειά σας αν εκλεγείτε συνενετικά εσείς. Να μου πείτε και εσείς τι θεωρείτε συνένεση μεταξύ των κυβερνήσεων. Πιστεύετε ότι η συνένεση μεταξύ υπηρεσιακή και μελλοντική κυβέρνηση θα σα δώσει περισσότερη δύναμη όσον αφορά το δύσκολο και δυσχερέ έργο σα. Απάντηση. Δεν θέλω να επιστρέφω σε αυτό το θέμα και να υποβληθώ σε ευκαιρία να στήσω, για να στήσω συγγνώμη αν προηγουμένως δεν εκφράστηκα σωστά. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη αν υπήρξε κάποια παρανόηση. Να πω ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από πολιτικές ε, συνενέσεις. Εμένα με πρότεινε μια κυβέρνηση ως υποψήφιο. Συνεπώς θεωρώ ότι η δύναμή μου για τον έλεγχο απορρέει ακριβώς από την θέση μου ως μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά παραλυπόμενα δεν με αφορούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κ. Σοντή. Μπορείτε να παραλάβετε την ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω εάν οι πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν σήμερα την Ισπανία αν ζητούσαν να αποσύρει την υποψηφιότητά το το δεχόταν γιατί στην δήλωσή του ε, λέει ότι αν υπήρχε αρνητική άποψη του, της Βουλής θα πέσυρε. Μα εγώ ερώτημα θέτω λέει ο Μιλόν. Οι πολιτικές δυνάμεις αν έλεγαν όχι, εγώ θέλω ας πούμε μια συνένεση την οποία επιθυμούν όλοι, την ευχόμεθα όλοι δεν θα είχαμε κανένα συμφέρον να έχουμε ε, κάποιον από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση να ελέγχει τους λογαριασμούς μιας δεξιάς κυβέρνησης στην Ισπανία. Λοιπόν, θα αποσύρατε την ε, υποψηφιότητά σας ενδεχομένως για να υπάρξει καλύτερη συμβαστική λύση. Εδώ υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Εγώ δεν υπέβαλα ποτέ υποψηφιότητα. Εγώ προσωπικά δεν υπέβαλα τίποτα. Με υπέβαλαν. και μέσω αυτή τη υποψηφιότητα είμαι εδώ. Χωρί την υποστήριξή σα, είναι δύσκολο να ασκήσω τα καθήκοντά μου στα πλαίσια του λεκτικού συνεδρίου. Δεν είχαν δείξει ούτε από την προηγούμενη ούτε από την τωρινή κυβέρνηση. Our Ωραία, η μας λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μόλις είδαμε ένα δανό υποψήφιο που προτάθηκε από μια κυβέρνηση η οποία ανέκυψε από πρόσφατες εκλογές και η πρότασή του ήταν απόλυτα θεμητή και νόμιμη κατά δική μας την άποψη. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την ίδια περίπτωση και για να μην πω και για τον Βέλγο υποψήφιο που έχουμε εδώ, ο οποίος ε, προέρχεται από μια μεταβατική κυβέρνηση, το ίδιο και ο κύριος Καλντέιρα, που τον πρότεινε μια κυβέρνηση, που και αυτή άλλαξε μετά τις εκλογές. Θεωρώ λοιπόν, εξάλλου είχα διαβούλευση με τις αρχές στη Μαδρίτη, οι οποίες κάνουν ακριβώς όλες τις αλλαγές. Είδα λοιπόν κατά πόσο ε, υπήρχε ε, πρόβλημα με την αντιπροσωπεία και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Λυπάμαι, Χριστίνα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να θίξω άλλο θέμα εδώ και να προσβάλλω κανένα, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία δεν αφορούν ούτε καν τι κυβερνήσει. Λοιπόν, σα ζητώ, όπω ακριβώ, όπω λέγει ο κ. Γάλια, σα ζητώ λοιπόν εδώ να αναλύσουμε και να εξετάσουμε υποψήφιου απόλυτα θεμητού από τις κυβερνήσεις. Εξετάσαμε τον Δανό, εξετάσαμε τον Βέλγο, μάλιστα η βελική κυβέρνηση είναι μεταβατική. Ε, δεν θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε υποψήφιο από το Βέλγιο επειδή έχουμε μεταβατική κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Και όπως είπε πολύ καλά και ο κύριος ε, Κορώνα, εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον να εκλεγεί ο κύριο ε, Κορώνα μετά από τι δικέ μου τι αποκαλύψει, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσω. Είναι ένας καλός επαγγελματίας, καλός τεχνοκράτη, ο οποίος προτάθηκε από μια νόμιμη κυβέρνηση όπως και άλλοι υποψήφοι και στο Κοινοβούλιο να μην αρχίσουμε να δημιουργούμε προηγούμενα. Αν ο κύριο Μούλτερ λοιπόν αποφασίσει να προτείνει κάτι άλλο, εγώ θα ακολουθήσω την ε, πρότασή του. Πάντω, θεωρώ ότι η δική μα Επιτροπή και γενικότερα το Κοινοβούλιο θα δημιούργησε ένα πολύ κακό προηγούμενο αν έκανε αναβολή, επειδή απλά και μόνο άλλαξαν οι κυβερνήσει στο ενδιάμεσο διάστημα τη υποβολή υποψηφιότητα. Δεν θα πρέπει εμεί να κάνουμε προσαρμογέ κάθε φορά που αλλάζουν ε, κυβερνήσει είχαμε τουλάχιστον άλλου δύο υποψήφιου, των οποίων η υποψηφιότητα προέρχεται από κυβερνήσει που είτε άλλαξαν είτε δεν έχουν αναλάβει τα καθήκοντά του. Θα ήθελα λοιπόν εμείς εδώ ως Επιτροπή να περιοριστούμε στην εξέταση του υποψηφίου που θεωρώ ότι έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα που ζητάμε και σήμερα το απόγευμα όταν καταλήξουμε στην απόφαση για την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου ή όχι να λάβουμε υπόψη και το διαδικαστικό θέμα. Όμως, ξαναλέω ότι δεν έχουμε μια κατάσταση μη νομιμότητας επειδή απλά και μόνο ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλους τους υποψήφιους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω λίγο πρόεδρος αυτά που είπε και προηγουμένως ότι εδώ συζητάμε τα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων και το απόγευμα θα συζητήσουμε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και θα ψηφίσουμε όλους τους υποψηφίους και ό,τι θέλουν οι βουλευτές. Τώρα όμως συζητάμε, αυτή είναι η πρόθεσή μας, τις τεχνικές, ε, τα τεχνικά προσόντα των υποψηφίων. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήλθατε στην Επιτροπή μας και θα συνεχίσουμε με τον επόμενο υποψήφιο σύντομα. I reopen and λοιπόν. λοιπόν, χαιρετίζω την κυρία Ιταλά και δεν ξέρω αν ανήκει ακόμα ήδη σε μας. Ε, σας δίνουμε Πέντε λεπτά όπως και σε όλους τους άλλους υποψηφίους για να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δέχεστε αυτή την υποψηφιότητα και τι εργασίες, τι ευθύνες θα αναλάβετε και τι τάσεις ε, όταν θα γίνετε ε, μέλος. Χαίρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πρέπει ωστόσο να ομολογήσω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε τέτοιου είδους ακρόαση σε αυτή την ωστή επιτροπή και είμαι λίγο νευρικός, ας το πούμε έτσι. Καταρχήν θα σας, πω, θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου. Ε, έχω γνωρίσει όλες τις κυβερνήσεις σε τοπικό επίπεδο, στην, στο δημοτικό, την πόλη Τούρκου, ε, σε κοινοβουλευτικό, στο κοινοβούλιο Είμαστε, ήμουνα μέλος της Συνταγματικής Επιτροπής, ε, δούλεψα στο Υπουργείο, στο Εσωτερικό, μαζί με τον Υπουργό και τώρα ε, ε, θέτω υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελεκτρικό, Ελεκτικό Συνέδριο. Πήρα μέρος σε πάρα πολλές ε, δικαστικές, είχα πάρα πολλά δικαστικά καθήκοντα, υπήρξα και ε, τον τελευταίο καιρό εκτός του ότι έκανα καράτε αλλά υπήρξα και εισαγγελέα. Είναι ένα ε, άθλημα το καράτε που μου έμαθε να σέβομαι τους αντιπάλους μου και να τους θεωρώ πραγματικά ίσους με μένα. Θέλω να σας πω δύο λόγια για το από πού προέρχομαι, για το παρελθόν μου ως ελεγκτής. Υπήρξα ελεγκτής για την Τράπεζα της Φιλανδίας και για την ε, φύτρα που είναι η ε, Τράπεζα Ανανέωσης της, της ε, Φιλανδίας. Επίσης δούλεψα για πάρα πολλές εταιρείες στα πλαίσια του Δήμου και έκανα, άσκησα έλεγχο και σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και ε, στις εταιρείες που συνεργαζόντουσαν με το Δήμο του Τούρκου. Πρέπει να πω ότι υπήρξα εισηγητής ε, ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αλλά όχι σε αυτήν την παρούσα επιτροπή. Αν εκλεγώ θα στραφώ θα εστιαστώ στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη συνεργασία. Αυτά θα είναι τα τρία κύρια σημεία που θα με απασχολήσουν. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη. Καταρχήν πρέπει νομίζω να αναρωτηθούμε, ο καθένας μας να αναρωτηθεί τι πρακτικές χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους μας και ασκούμε ε, μία αξιολόγηση κριτική της εργασίας μας ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία για να ξέρουμε, να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς πετυχαίνουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Πέρα από αυτό πιστεύουμε ότι είναι ε, ο έλεγχος ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αποδεικνύεται πώς έγιναν οι δαπάνες, αν έγιναν σωστά και αν υπάρχει πρόοδος ή αν δεν υπάρχει καμία πρόοδος υπάρχει, είμαστε πολύ μακριά από το στόχο μας ε, για την ώρα αλλά είχαμε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια και μπορούμε να πούμε σήμερα ότι τα όσα διαθέτουμε δεν είναι αρκετά. Πρέπει να βρούμε μια λύση για το πώς θα ελαχιστοποιήσουμε το περιθώριο λάθους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έπρεπε να ασκεί κυρώσεις στα κράτη-μέλη. Ύστερα η διαφάνεια είναι ένας ε, ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε πώς έχουν δαπανηθεί τα χρήματα. Πέρα από αυτό ε, πρέπει να πληροφορούμε τους ε, φορολογουμένους και τους πολίτες και όλοι να έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση, πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε όλη την τεκμηρίωση που χρειάζεται για να μπορεί να γίνεται η σωστή κρίση των ε, ικανοτήτων του συνεδρίου. Ο τρίτος στόχος μου είναι η συνεργασία κύριε Πρόεδρε και ειδικά με τα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό πρέπει να βρούμε ένα πνεύμα συνεργασίας και κοινών στόχων με όλους. Ο καθένας μας πρέπει να δεσμευτεί ως προς αυτό. Στη σημερινή κρίση είναι υψής της σημασίας να δαπανώνται σωστά οι πόροι που διαθέτουμε. Και εδώ πιστεύω ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σοβαρό κρίσιμο ρόλο. Είναι λοιπόν για μένα εξαιρετική σημασία να πάρω μέρος σε αυτή την εργασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και κατά τη συνήθειά μας δίνω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ιτάλα Η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει αυτή η δραστηριότητά σας για το καράτε και άλλες δραστηριότητες που έχετε, αστυνομικές κλπ. Εκτός από τις τρεις αρχές που αναφέρατε, πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο, που καταδεικνύουν την ικανότητα και την τιμιότητά σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Όταν έρθετε από την άλλη μεριά, στο αγγλικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό δηλαδή, με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να διακυπεραιώσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ή τις αλλαγές που χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό. Για το βιογραφικό σας να αναφέρω επίσης κάποιες αμφιβολίες ή κάποιες απορίες που έχω Λέτε ότι είστε αναπληρωτής αστυνομικό διοικητή, αναπληρωτή δικαστικό αναπληρωτής δικαστικός αστυνομικό αναπληρωτής αστυνομικός Δεν ξέρω αν είναι η μετάφραση λανθασμένη ή πώς ακριβώς ήταν η πω ακριβω ηταν η θέση σα. Είπατε επίσης ότι εσείς θα εγκαταλείψετε όλες τις δραστηριότητες σας στη Φιλανδία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν διοριστείτε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Πώς θα το κάνετε αυτό, ευχαριστώ. Κύριε Τάλα, αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγκεντρία για τις ερωτήσεις της. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι μπορώ να σας μεταβιβάσω όλα όσα έχω διδαχθεί ως μέλος της Επιτροπής. Θα ήθελα να συμβάλλω με τις εμπειρίες μου στο ελεγκτικό συνέδριο και να επηρεάσω με την εμπειρία μου τις εργασίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω εργαστεί εδώ επί και θεωρώ ότι η τρέχουσα σύνθεση του ελεγκτικού συνεδρίου διασφαλίζει ότι τα διάφορα άτομα με τις διαφορετικές τους εμπειρίες και το διαφορετικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο μπορούν να συνεργαστούν και σε αυτό το πλαίσιο θα θέλω να συνδράμω. Σε ό,τι αφορά τις αντιπροσωπείες στον τομέα της αστυνομία. θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν ήταν ε, σταθερή η θέση μου, απλά για μικρά και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ανέλαβα τα καθήκοντα αυτά. Για παράδειγμα, όταν ε, έλειπε κάποιος σε διακοπές ή για άλλους λόγους. Ανέλαβα λοιπόν τα καθήκοντα αυτά και συνέλεξα μεγάλες εμπειρίες ε, στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποχρεώσεις μου. Στις διάφορες επιχειρήσεις ε, στις οποίες συμμετείχα μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι σαφές ότι προφανώς θα σταματήσω τις δραστηριότητε αυτές μόλις εκλεχθώ στο ε, ε, ελεκτικό συνέδριο. Κυρία Ιβάνοβα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ήταλα. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, καλωσορίσω εδώ. Χαίρομαι που βρίσκεστε μαζί μας και που μας μιλάτε και είστε ένας από τους λίγους υποψήφιους που τόνισαν πόσο σκοπεύουν να συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοκομπού. Άρα υπολογίζουμε σε αυτό. Έχω θέσει το ίδιο ερώτημα και σε άλλους υποψηφίους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των χρηματοοικονομικών μέσων. Πώς θεωρείτε ότι διαμορφώνεται ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση την αποδοτικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το EFSM. Με 60 δις ευρωπαϊκούς πόρους που θα το διαδεχτεί το ESM το 2013. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στη συνθήκη προς το παρόν για το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Τι θα κάνετε όμως για να διασφαλίσετε ότι θα δραματίσει ενεργό ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Σίταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ελεγκτικό συνέδριο στην παρούσα χρονική συγκυρία. Βρισκόμαστε σε μια φάση πολύ σοβαρή κρίση και μάλιστα δεν διαφαίνεται καν το τέλο της κρίση. Ξεκινήσαμε λοιπόν στα πλαίσια της κρίση να διαμορφώνουμε μηχανισμούς για την σταθεροποίηση και για την διάσωση. Και φυσικά οι πολίτες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι βέβαιοι για τη λειτουργία των μέσων αυτών. Θεωρώ ότι μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά, αλλά μιλάμε και για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου ο μηχανισμός, ο μηχανισμός ελέγχου θα πρέπει να είναι εξαιρετικά αξιόπιστος. Αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα, θα πρέπει με τον βέλτιστο τρόπο να διεξάγει αποτελεσματικούς ελέγχους και να έχει όλα τα μέσα που χρειάζεται στη διάθεσή του προκειμένου να ασκείται και κοινοβουλευτικό έλεγχος ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός. Θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη όταν μιλάμε για τόσο τεράστια χρηματικά ποσά. Και εδώ είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια στην ε, χρήση των μέσων. Ο ρόλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου ασφαλώς και θα αλλάξει στο μέλλον σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αυτό. Ο κύριος Ροντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά να πω το πόσο χαίρομαι που οι χώρες ή οι κυβερνήσεις επιλέγουν προσωπικότητες για την άσκηση καθηκόντων σε οργανισμούς όπως το Λευκό Συνέδριο αυτό είναι ένα σημάδι ποιότητας και να πω στον συνάδελφο ότι χαίρομαι πολύ που επιλέχθηκε και να το πω επίσης ότι εκτίμησα πολύ τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και ιδιαίτερα στο θέμα των επαφών με τα εθνικά λεκτικά συνέδρια. Θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ελπίζω μελλοντικό μέλος του Ευρωπαϊκού Λεκτικού Συνεδρίου. Συχνά συζητάμε το πολιτικό ή το τεχνοκρατικό προφίλ και ο υποψήφιος που έχουμε μπροστά μας τώρα είχε ένα σημαντικό παρελθόν κυβερνητικών θέσεων και ευθυνών και ταυτόχρονα έχει και τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και προσόντα κάτι το οποίο νομίζω θα έκανε ένα πολύ καλό μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου και το οποίο χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε ή όχι. Έχετε το λόγο όπως και να έχει. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, να προσθέσω κάτι. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία ασφαλώς αποτελούν σημαντικές αρχές. Ωστόσο, η συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να βρούμε από κοινού και στα μάτια των πολιτών να είμαστε αξιόπιστοι. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πέρα από, την, ε, από τον έλεγχο του προϋπολογισμού και εργασίες άλλων επιτροπών. Μιλάμε για παράδειγμα σήμερα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση της ε, αγροτικής πολιτικής. Είναι πολύ σύνθετο το εγχείρημα αυτό και θεωρώ ότι κατά την φάση κατάρτιση της νομοθεσίας αυτής θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των σχετικών ταπαντών που θα προκύψουν. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο είναι κάτι το αναπόφευκτο. Υπάρχουν πολλοί τομεί συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, η κυρία Γκρέσλε. Αγαπητέ Βίλε, ελπίζω ότι θα καταφέρει να μειώσει την απόσταση μεταξύ ε, Λουξεμβούργου και Βρυξελών. Ε, αυτό προσδοκούμε. Έκκληση δική μου για τις ειδικέ εκθέσεις να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο που να αξίζουν τον κόπο, γιατί υπάρχουν δύο αντιφατικά στοιχεία με την Επιτροπή και στο εσωτερικό του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν ξέρω τι θα απομείνει. Αλλά αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί αν συνεχίσει το ελεγκτικό συνέδριο όπως ε, συνεχίζει σήμερα ανακύπτουν άλλα ζητήματα. Ασχολήθηκα με τους ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς και τις αντιρρήσεις των κρατών μελών. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε σαφή λόγια, να μιλάμε μια σαφή γλώσσα. Θέλουμε λοιπόν συντομία και συνοπτικότητα στις εκθέσεις αυτές. Γι' αυτό λοιπόν η έκκλησή μας για συνεργασία. Το θέμα είναι λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται για τον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι όμως αστείο. Θέλουμε μία φιλική συνεργασία. Γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ το ελεγκτικό συνέδριο για να αποκαταστήσουμε το έλλειμμα εμπιστοσύνη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ήτελα έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας. Μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ε, κρατών μελών θα πρέπει να υπάρχουν πιο καλές σχέσεις, πιο στενές σχέσεις. Και στο παρελθόν έχω βιώσει το πόσο προβληματικές μπορεί να είναι αυτές οι σχέσεις. Ελπίζω λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να συντάσει πιο επίκαιρες εκθέσεις. Προκειμένου να εξετάζουμε θέματα που απασχολούν τον πολίτη. Προκειμένου να ξανακερδίσουμε την χαμένη εμπιστοσύνη. Έχω μακρά εμπειρία με τη σύνταξη εκθέσεων και ξέρω ποια προβλήματα ανακύπτουν και σε ό,τι αφορά ζητήματα κατανόησης. Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι οι εκθέσεις θα πρέπει να καταστούν πιο αντικειμενικές. και γι' αυτό θα ήθελα να συμβάλλω στην άρση των αδυναμιών, προκειμένου να καταστούν πιο επίκαιρε και πιο κατανοητέ οι εκθέσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητά κανεί άλλο το λόγο. Άρα, ο λόγο και πάλι στην εισηγήτρια για να συνοψίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω στην συνάδελφο Ιγκεμπόρκ ότι δεν θέλουμε να υποβοηθά εμά, θα πρέπει να είναι εξάρτητο και από το Κοινοβούλιο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η συνάντηση προηγουμένω για Κορτίνε που λείπει τώρα, νομίζω ότι οδήγησε στην παρανόηση ότι ο καθένα ορίζει το δικό του μέλο στο ελεκτικό συνέδριο. Δεν είναι έτσι και ελπίζω να μην είναι έτσι. Ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Ήταλα για τις απαντήσεις του και κυρίως για την δημιουργική του ικανότητα αυτή τη στιγμή άγχους γιατί η διάδοση των εκθέσεων της Επιτροπής μας σε άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι καλή ιδέα. Δεν ξέρω αν το επιτρέπουν αυτό οι πόροι που διαθέτουμε, αλλά είναι από μόνη της καλή ιδέα. Ώστε να υπάρχει μέσω ανεξαρτησία, συνεργασία και να κερδίσουμε και τους πολίτες και την κοινή γνώμη. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά και νομίζω ότι σε περίπτωση που εσεί είστε, κύριε Ιταλά, μέλο του Λεκτικού Συνεδρίου, θα έχουμε ένα θαυμάσιο επιχείρημα στο όργανο αυτό για να πετύχουμε την αναθεώρησή του και την σωστή του λειτουργία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται η πρένη μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ήταλα και ελπίζω να τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα με όλους σας. η κυρία Κρέσλε, θα ήθελα να παραπονεθώ για την ε, θερμοκρασία στην αίθουσα, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Θα το φροντίσουμε, λέει ο πρόεδρος. <laughs>